Hello. Welcome everybody. Χαίρετε. Ε, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Ίσως να, να προεδρεύσω σήμερα. Καλώς ήρθατε και καλωσορίζουμε μία αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν που θα παρακολουθήσουν ένα τμήμα των εργασιών μας. Είναι πολύ σημαντικό που ε, θα παρακολουθήσετε τις εργασίες της Επιτροπής ε, Γυναικών. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Χαιρετίζω τους προσκεκλημένους μας από το Αφγανιστάν, μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια και βεβαίως ε, έχει δεσμευθεί το Αφγανιστάν να εδραιώσει τη δημοκρατία και να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών. Ένα πρώτο θέμα που είναι πολύ σημαντικό και που το έχουμε ήδη συζητήσει είναι η εξάλληψη του ακροτηριασμού των γενετικών οργάνων των γυναικών. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για αυτό το θέμα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που περιέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Γιατί είναι δύσκολο να συλλεγούν αυτά τα στοιχεία Είναι εδώ λοιπόν η έκθεση, εδώ έχουμε αντίγραφα στη διάθεσή σας. Τώρα είναι η συνεδρίασή μας ε, με ανοιχτή διαδικασία. Πρώτα θα, πάρει, θα πάρουν το λόγο οι προσκεκλημένοι μας, μετά θα πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά, γι' αυτό ακριβώς ανοιχτή διαδικασία, θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο όχι μόνο οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές, αλλά και όσοι από, τις, από τους παρευρισκόμενους επιθυμούν να παρέμβουν. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να παρέμβουν όσοι το επιθυμούν. Ο πρώτος μας ε, προσκεκλισμένος είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια χώρα που είναι ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυτό, είναι η κυρία Νάνα Οτού Ογιόρτε. που έχει μεγάλη εμπειρία για τα θέματα αυτά του ακροτηριασμού των γυναικείων γενικών οργάνων είναι εκτελεστικός διευθυντής του Forward που είναι στην πρωτοπορία της ε, αντιμετώπισης του θέματος αυτού στον Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει πολλή δουλειά για το θέμα αυτό αλλά όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν πως ήταν Ε, χαιρόμαστε λοιπόν που η κυρία, η κυρία ε, ο, έχει το λόγο ε, για να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Μας είπε ότι θα μας παρουσιάσει και μερικά πολύ διαφωτιστικά βίντεο η κυρία Νάννα, έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων που έχω τη δυνατότητα σήμερα να βρίσκομαι εδώ και να σας μιλήσω για την προστασία των κοριτσιών από ε, τον γενετήσιο ακροτηριασμό. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια προβολή που θα ε, διαρκέσει τρία λεπτά.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 we can end FGM. This is a traumatic experience. Πρόκειται για τραυματική εμπειρία. Και όπως λέει και η Τενιούλα, μπορούμε μαζί να δώσουμε τέλος σε αυτή την πρακτική. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του, μαζί όμως μπορούμε. Εκπροσωπώ την οργάνωση Forward, που είναι ίδρυμα για τις ε, έρευνες ε, για την υγεία των γυναικών. Το 1985 ιδρυθήκαμε και δραστηριοποιούμαστε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και σε τέσσερις χώρες της Αφρικής επικεντρωνόμαστε κυρίως στον γενετήσιο ακροτηριασμό των γυναικών, την, τους γάμους μεταξύ παιδιών και... Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας έχει να κάνει με τον γενετήσιο ακροτηριασμό γυναικών. Καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχει πολλή σχέση ανάμεσα στα τρία αυτά θέματα. Το μευτικό συρίγγιο και ε, τον ακροτηριασμό των γυναικών και τους ε, γάμους μεταξύ παιδιών. Τα θέματα που συζητάμε ε, είναι παγκόσμια. Ε, ξέρουμε ότι ο ακροτηριασμός γυναικών ε, γίνεται όχι μόνο στην Αφρική, αλλά σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί κάποια μορφή ακροτηριασμού και κάποιες νέες μελέτες του ΟΗΕ επιβεβαιώνουν τα στοιχεία. Όσον αφορά τους γάμους μεταξύ παιδιών, ένα στα έξι κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών είναι ήδη παντρεμένα ή συγκατοικούν υπό κάποια τέτοια μορφή. Και επίσης το 75% ε, των ε, γυναικών ε, με, με ε, είχαν γένα που διήρκησε πάνω από 3-24 ώρα. Θα μιλήσω λοιπόν για τη δουλειά της οργάνωσής μας ε, και Επειδή είμαστε οργάνωση γυναικών ε, της ε, Αφρικανικής Διασποράς, πιστεύουμε ότι χρειάζεται να έχουμε μία φωνή, διότι είναι θέματα αυτά που μας αγγίζουν βαθιά. Και ε, μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη πολιτικής και η και πρακτικών σε τι στρατηγικά επίπεδα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου έχουμε αρκετά μεγάλη κοινότητα. Πολλούν, ε, έχουν μεταναστε... Πολλές ε, γυναίκες έχουν μεταναστεύσει εκεί από την Αφρική. Στην Αφρική είναι πιο έντονα τα προβλήματα. Και θέλουμε επίσης να συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η δουλειά μας ε, λοιπόν ε, σε αυτά τα τρία επίπεδα είναι απαραίτητη και η ανάπτυξη πολιτικών ε, σημαίνει ότι πρέπει να Είμαστε δραστήριοι όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Αφρική και στην Ευρώπη γενικά, σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου Εξετάζουμε τέσσερις τομείς ε, συμβουλές ε, προς τους νέους ε, και συμμετοχή των νέων, να επιτρέπουμε στους νέους να προστατεύονται. με τη δουλειά τους, με τους συνομήλικους τους, αλλά και με την πρόσβαση σε, στις απαραίτητες υπηρεσίες. Το επιτρέπουμε αυτό. Τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε πονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγέ ε, και ε, επιτρέπει να ακουστεί η φωνή των νέων. Επίσης έχουμε κατάρτιση ε, επαγγελματιών που τους επιτρέπει να έχουν τις δεξιότητες και τη γνώση για να ανταποκριθούν σωστά όταν συναντούν κορίτσια και γυναίκες που έχουν υποστεί γενετήσιο ακροτηριασμό. Το πρόγραμμά μας στόχο έχει να διασφαλίσει τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών οι οποίοι να προστατήσουν ώστε να έχουμε βιώσιμη αλλαγή, να έχουμε μία μόνιμη αλλαγή της κατάστασης. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με συμβούλους υγείας σε τοπικό επίπεδο και με άλλους παράγοντες σε τοπικό επίπεδο. Η δουλειά μας λοιπόν, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής, συνδέεται με τη διαμόρφωση πολιτικής όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και πιο συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εργασίε μα βασίζονται σε έρευνε και θα ήθελα να σα δώσω κάποια στοιχεία από έρευνε που κάναμε στο Λονδίνο. Είχαμε μία έρευνα που δείχνει τι λένε οι ίδιες οι κοινότητες. Μία κυρία από το Κουρδιστάν έλεγε ότι ε, οι άνθρωποι δεν συζητούν το θέμα του γενετήσιου ακροτηριασμού των γυναικών. Στο παρελθόν κανεί δεν συζητούσε το θέμα αυτό. Μία κυρία από την ε, Γκάμπια είπε ότι πάντα υπάρχουν διαφορέ ε, απόψεων. Μερικοί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνεται και άλλοι λένε όχι. Δεν είναι θέμα θρησκευτικό, είναι θέμα πολιτιστικό. Μία νέα γυναίκα από τη Σιέρα Λεόνε είπε ότι στην κοινότητα Μπούντου, ε, εάν ε, υποστεί κανείς γενετήσιο ακροτηριασμό, ε, θα έχει κανείς τον σεβασμό των άλλων. Και άλλη μία γυναίκα από την Κάμπια είπε ότι επέστρεψα στην Κάμπια με τα παιδιά μου και είδα την οικογένειά μου. Ε, η μητέρα μου ήθελε ε, τα παιδιά μου να υποστούν ε, γενετήσιο ακροτηριασμό και της είπα ότι θα με βάλουν φυλακή στο Ηνωμένο Βασίλειο αν το επιτρέψω. Οπότε είπε εντάξει τότε άστο. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τις φωνές των κοινοτήτων για να πετύχουμε αποτελέσματα και να συνεργαστούμε με αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική. Ο νόμος ε, είναι καθοριστικής σημασίας. Ε, παρότι φαίνεται να μην λειτουργεί, παρόλα αυτά είναι ένας ε, παράγοντας προστασίας. Πολλές γυναίκες το χρησιμοποιούν αυτό ως εργαλείο όταν επιστρέφουν στις πατρίδες τους δουλειά που κάναμε στον Πρίστολ βασίστηκε στις έρευνες αυτές μεταξύ των γυναικών των ε, διαφόρων ε, αφρικανικών κοινοτήτων και έτσι τώρα στο Πρίστολ με βάση τις έρευνες ε, έχουν διαμορφωθεί διάφορες πολιτικές και πρακτικές σε επίπεδο πόλης. Η δουλειά με τους νέους συμπεριλαμβάνει δουλειά στα σχολεία. Η δουλειά που κάνουμε εκεί βασίζεται σε ένα μοντέλο που ονομάζεται το Χρυσό Τρίγωνο. Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία, με το προσωπικό των σχολείων συνεργαζόμαστε. η δουλειά μας απευθείας, που απευθύνεται απευθείας στους ε, ανθρώπους και ε, ε, στους μαθητές και στους γονείς. Η δουλειά που γίνεται στα σχολεία θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αποφυγής βλάβης, να υπάρχει μια ασφαλής περιοχή στα σχολεία, να υπάρχει ασφαλές περιβάλλον για όλους, αλλά να υπάρχει και ενημέρωση σχετικά με τον γενετήσιο ακροτηριασμό στην σχολική ύλη και να υπάρχει ενημέρωση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πρακτικοί παράγοντες. Πάνω απ' όλα όμως η δουλειά στα σχολεία στόχο έχει την ενδυνάμωση και συμμετοχή των νέων. το σχολικό μας πρόγραμμα με την υποστήριξη της κυβέρνησης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πετύχει καλά αποτελέσματα. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στην ανάγκη να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ των χωρών. Ο γενετήσιος ακροτηριασμός των γυναικών είναι ένα πρόβλημα ε, διεθνές και απαιτεί και διεθνείς λύσεις, ε, το να οικοδομήσουμε γέφυρε ε, ε, προς τις χώρες προέλευσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε στην Ευρώπη να εργαστούμε απομονωμένοι πάνω στο θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διάλογο με χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε οργανώσεις πολιτών να παρέχουμε ε, συμβουλές και χρηματοδότηση και να επιτρέπουμε στις ε, τοπικές οργανώσεις ε, να αναπτύσσονται. Θέματα όπως η γάμη μεταξύ παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών είναι θέματα για τα οποία θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση για να πετύχουμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Θα ήθελα να αναφερθώ και στις ε, εταιρικέ ε, σχέσεις ε, που έχουμε οικοδομήσει. Στο πλαίσιο αυτών έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε γέφυρες στην Ευρώπη. Η οργάνωση Forward είναι μέλος του δικτύου End που στόχο έχει την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων. Έχουμε 19 μέλη από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργαζόμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του γενετησίου ακροτηριασμού γυναικών στην Ευρώπη. Ε, τον επόμενο μήνα θα, εκδοθεί, θα δημοσιευτεί η έκθεσή μας, την οποία έχω εδώ, που προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τις ε, οργανώσεις της κοινωνίας ε, των πολιτών. Έχουμε πετύχει καλά αποτελέσματα προεδρεύοντας σε συνοργάνωση αυτή. Ε, είμαστε ευγνώμονες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτρέψει στο δίκτυο αυτό με χρηματοδότηση και υποστήριξη ε, να αναπτυχθεί περαιτέρω. Μια άλλη εταιρική σχέση που έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε στην οργάνωση Forward είναι με την Αφρική. Η οργάνωση Forward συμμετέχει στην ε, κοινοπραξία Girl Generation. Είμαστε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που ε, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 υπό την ηγεσία του Αρτόκανο που πρωτοστάτησε στην ε, ε, εξάλληψη του γενετήσιου ακροτηριασμού. Έχουμε το κοινό πρόγραμμα UNICEF UNFPA ε, καθώς και το πρόγραμμα ερευνών που συλλέγει στοιχεία. Προσπαθούμε λοιπόν να πετύχουμε κοινή κατανόηση και συνεργασία για να πετύχουμε την εξάλληψη του γενετήσιου ακροτηριασμού. Συχνά στην Αφρική όσοι δουλεύουν πάνω στο θέμα αυτό δουλεύουν απομονωμένοι. Θέλουμε λοιπόν να συντονίσουμε τις προσπάθειές τους. Επίσης, ε, ένα θέμα που έχει παραμεληθεί στο θέμα αυτό είναι η συνεργασία με τους άντρες. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα Men Speak Out, που είναι το πιο στρατηγικό μας πρόγραμμα, και έχουμε εταίρους στο Βέλγιο και τις κάτω χώρες ε, και στόχο έχει το πρόγραμμα να ακουστεί η φωνή και των ανδρών ώστε να παίξουν και οι άνδρες ε, στρατηγικό ρόλο ε, στην εξάλληψη της πρακτικής αυτής. Επίσης, ασχολούμαστε με την κατάρτιση, συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα γνώσης της Ευρώπης, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήθελα να τονίσω και τη σημασία ε, Τη σχέση ε, του γενετήσιου ακροτηριασμού με άλλα θέματα, όπως είναι ο γάμος μεταξύ παιδιών. Σε πολλές χώρες ε, συνδέονται τα δύο αυτά θέματα στενά μεταξύ τους. Σε άλλες χώρες συνδέεται και με τους, με τους καταναγκαστικούς γάμους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του γενετήσιου ακροτηριασμού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις. Συχνά δεν έχουμε αποδείξεις ε, για το ποιες λύσεις λειτουργούν καλύτερα. Ε, ο γενετήσιος ακροτηριασμός δεν περιορίζεται στην Αφρική, ε, πραγματοποιείται και στην Ασία και στην Μέση Ανατολή και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις χώρες αυτές. Υπάρχει πολύ λίγη υποστήριξη από ειδικού ε, και δεν υπάρχει στρατηγική χρηματοδότηση για ε, ε, παρεμβάσεις εντός των κοινοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι για να πετύχουμε πρόοδο θα πρέπει να συνεργαστούμε. Και θα ήθελα να κλείσω με μια πιο θετική ταινία πάνω στον γενετήσιο ακροτηριασμό που δείχνει την ε, πραγματική ιστορία της Κάτι και Ρώτη.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 Thank you very much. It's been a pleasure talking to you about Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά μου να σας μιλήσω για τη δουλειά μας ε, και ε, που βλέπω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά εάν συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ότο Γιορτέη, ιδίως για το ευτυχές αυτό τέλος που είχε η δεύτερη ταινία που μας δείξατε, όντως πραγματικά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αν συνεργαστούμε. Ας απευθυνθούμε τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Ότο Γιορτέ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίασή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την παραβίαση αυτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των παιδιών και η δέσμευσή μας φαίνεται και από την ανακοίνωση του 2013 για την εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς επίσης και στη στρατηγική μας δέσμευση για την ισότητα των φύλων από μια βιασική δράση είναι η εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στα πλαίσια της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Αντιλαμβάνουμε δράση πολύ γρήγορα σε τρία σημεία. Πρώτον, βελτίωση της γνώσης και συγκέντρωση πληροφοριών. Δεύτερον, δράσεις πρόληψης, προστασίας, ποινική δίωξη και εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων παγκοσμίω. Θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα λίγο περισσότερο στα δεδομένα και στην συγκέντρωση των δεδομένων αυτών και στην γνώση που απορρέει από τα δεδομένα αυτά. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι φαίνεται, περίπου 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίω έχουν υποστεί γενετήσιο ακροτηριασμό και ένα μισό, μισό εκατομμύριο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για αρχικές μόνο εκτιμήσεις, δεν έχουμε επίσημα στατιστικά δεδομένα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κλίμακα της εμφάνισης του φαινομένου αυτού. Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μια εκτίμηση των κοριτσιών που κινδυνεύουν από γενετήσιο ακροτηριασμό και δεν έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίε για το πού γίνεται ο ακροτηριασμό αυτό και από ποιου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη συλλογή των δεδομένων. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε εσεί επίση στη μελέτη που κάνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, όπου και εκεί έχουμε κάποιε εκτιμήσει. Έγινε μια πιλωτική δράση σε τρία κράτη-μέλη και τα επόμενα χρόνια, μάλλον του χρόνου, θα έχουμε πέντε ακόμα κράτη-μέλη τα οποία θα ενταχθούν σε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα στην ανάλυση αυτή που κάνει το Ευρωπαϊκό Αυτό Ινστιτούτο. Έγινε επίση και μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο τη Γκέντα προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια κοινή μεθοδολογία όσον αφορά την εμφάνιση, τη συχνότητα μάλλον τη εμφάνιση του φαινομένου αυτού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Στα πλαίσια τη ανακοίνωσή μα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται πάρα πολύ στο ζήτημα τη πρόληψη. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια βιώσιμη κοινωνική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτούμε εθνικές εκστρατείες, αλλά επίσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε διάφορα διεθνικά προγράμματα που προσπαθούν επιτόπου να επιφέρουν πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών. Ένα από τα πράγματα που θέλω να τονίσω είναι τα πιλωτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία θα είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες εκείνους που είναι σε άμεση επαφή με κορίτσια τα οποία κινδυνεύουν ή με θύματα γενετήσιου ακροτηριασμού και αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε διδάσκοντες, καθηγητές, αστυνομικούς, νοσοκόμες, δικηγόρους κτλ. Ελπίζουμε ήδη από το χρόνο να έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις για το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα διαρκέσει δύο χρόνια και έχει επιτευχθεί χάρη στα πιλωτικά προγράμματα τα οποία πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την ποινική δίωξη, να επιστήσω την προσοχή σας σε μία ανάλυση η οποία δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2016 όσον αφορά τι δικαστικές υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το γενετήσιο εκροτηριασμό, προσπαθήσαμε να δούμε τι έχει γίνει στα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν καταφέρει να προχωρήσουν με ποινικέ τέτοιε διώξεις άλλα πάλι όχι. Και από εκεί όμω μπορούμε να δείσουμε κάποια διδάγματα. Έχουμε έπειτα τη διεθνή προστασία. Έχουμε εδώ πέρα μία αναδιατύπωση της ε, οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου Ξέρετε ότι και στα πλαίσια της οδηγίας αυτής θα πρέπει να καλυφθούν, ήδη καλύπτονται μάλλον, οι γυναίκες αυτές οι οποίες κινδυνεύουν από γενετήσιο ακροτηριασμό, προτείνονται κάποια ελάχιστα πρότυπα και επίσης στα πλαίσια της εξωτερικής της δράσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει σε συνεργασία που έχει με τρίτες χώρες να προωθήσει και τον πολιτικό διάλογο και το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δράσει κατά του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία ήθελα να θίξω στην παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And now it's time for... Ευχαριστώ. Και τώρα μπορείτε να πάρετε το λόγο. Όλοι όσοι είναι στην αίθουσα μπορούν, να θέλουν, να πάρουν το λόγο. Όπως σας είπα, μπορούν όχι μόνο οι ευρωβουλευτές, αλλά όλοι οι παρευρισκόμενοι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις ή να κάνουν συστάσεις. Και έχει δει το λόγο η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στο Bristol, γιατί έχετε εδώ δύο ευρωβουλευτές από την περιοχή και ξέρω τι καλή δουλειά κάνετε εκεί. Καταπληκτική. Έχω ορισμένε ερωτήσεις. Πρώτη, όταν ε, συζητούμε με τις ακτιβίστρες στο Bristol, μας είπαν ε, κάτι που έχει ενδιαφέρον. Τα ταξίδια που κάνουν ε, τα νέα κορίτσια. Δεν ξέρω αν ε, προσπαθείτε να δείτε από τον τρόπο με τον οποίο τη συχνότητα και τους προορισμούς μπορείτε να καταλάβετε τι επίκειται να γίνει ή θα μπορούσαμε να παρέμβουμε σε άλλα στάδια της διαδικασίας. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το πώς ασκείται δίωξη ή πώς εφαρμόζεται ο νόμος για τους ακροτηριασμούς. Ναι, μεν εφαρμόζεται ατελώς, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει νόμος είναι κάτι που μπορούν να το οι γυναίκες να πούν ότι δεν το κάνω γιατί φοβάμαι ότι θα διωχθώ. Αλλά θέτε θέματα γι' αυτό και για να αντιδράσω και σε αυτό που μόλις είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα έπρεπε να γίνονται οι διώξεις και πώς γίνονται και ποιοι θα πρέπει να διώκονται. Και τέλος η προφανής ερώτηση. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τι άλλα θέματα θα μπορούσαμε να προωθήσουμε. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν θέματα με τα ταξίδια, με τις μετακινήσεις. Το καλοκαίρι, όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, πρέπει να δημιουργούμε περισσότερο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό. Το... Στον Πρίστολ, ε, στην αρχή του καλοκαιριού, ξεκινήσαμε μια καμπάνια. Και επίσης πρέπει να συζητάμε και στους προορισμούς με γιατρούς και νοσοκόμες αλλά δεν φαίνεται οι γιατροί και νοσοκόμες να είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι γιατί κάποιες τοπικές αρχές προσπαθούν να εκπαιδεύσουν αλλά ορισμένες εκπαιδεύσεις είναι μόνο αποσπασματικές οπότε δεν είναι αρκετά καταρτισμένοι ορισμένοι επαγγελματίες της υγείας για να ξεκινήσουν μια συζήτηση για το θέμα αυτό ένα άλλο θέμα σε σχέση με τα ταξίδια Πρέπει να συμμετέχουν ευρύτερα οι κοινότητες. Δεν έχουν γίνει καμπάνιες ε, που να απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινότητα λίγο πριν το καλοκαίρι, παρά το ότι ήταν σύσταση αυτό της Επιτροπής του Ηνωμένο Βασίλειο του Υπουργείου Εσωτερικών για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν έγινε τέτοια εκστρατεία. Οπότε οι συζητήσεις αυτές, ε, οι συζητήσεις στην κοινότητα θα ευαισθητοποιήσουν τις κοινότητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα για τις διώξεις. Σε πολλές κοινότητες ακούμε ότι όσοι έχουν εμπλακεί με το πώς λειτουργεί ο νόμος, όσοι δηλαδή είναι επαγγελματίε στον κλάδο αυτό, ξέρουν να τον εφαρμόσουν. Αλλά πρέπει λοιπόν να μάθει ευρύτερα η κοινότητα ποιος είναι ο νόμος και ποιες θα είναι οι ποινές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και στον Bristol για παράδειγμα, έγινε μια καταγγελία και παρόλα αυτά η μητέρα πήρε τα παιδιά της και μπόρεσε να ταξιδέψει παρά το ότι υπήρξε καταγγελία ότι θα ακροτριαστούν στον προορισμό που θα πήγαιναν. Είναι σαφές λοιπόν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταδικαστεί κανένας. Καμία οικογένεια δεν έχει καταδικαστεί γιατί υπέβαλε τα παιδιά της, τα κορίτσια της σε αυτόν τον ακροτηριασμό. Αλλά ακόμη και συζήτηση για τον νόμο βοηθάει. Ναι, στη Γαλλία έγιναν περισσότερες διώξεις. Αλλά ακόμη και στη Γαλλία κινδυνεύουν τα κορίτσια. Ναι, οι διώξει είναι ένα στοιχείο μιας στρατηγικής. Αλλά πρέπει να υπάρξουν και άλλες στρατηγικές πρόληψεις, να δουλέψουμε στα σχολεία, στις κοινότητες και πάνω απ' όλα να δεσμευτούμε και με τις κοινότητες προέλευσης. Και πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι η χρηματοδότηση δίνεται μόνο για δράσεις στην Ευρώπη και όχι στην Αφρική. Άρα το βασικό είναι και οι κοινότητες στις χώρες προέλευσης να ενημερωθούν. Εάν δεν υπάρχουν οργανώσεις που να μπορούν να παρακολουθήσουν πού ακριβώς πάνε όσοι επιστρέφουν στην Αφρική, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τις αναγκαίες δομές και στα δύο μέρη. δουλειά μόνο στην Ευρώπη δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να δράσουμε και στην Αφρική με συμμετοχή και κοινοβουλευτικών εκεί για να γίνει περισσότερος διάλογος για να διασφαλίσουμε ότι το θέμα αυτό θα είναι στην επικαιρότητα και θα συζητιέται σε βάθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρλινγκ ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας όπως ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες και οι προβολές που είδαμε. Ιδιαίτερα η πρώτη, νομίζω θα έπρεπε να αποτελεί υποχρεωτική ύλη στα σχολεία από μια ηλικία και μετά. Όπως και η Κλέρ και εγώ, χάρηκα που αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο Μπρίστολ. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο θέμα της δίωξης, της ποινικής δίωξης, διότι Ξέρουμε ότι κάποια κρατημέλη έχουν υψηλότερα επίπεδα και από ό,τι κατάλαβα, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ε, τα νούμερα μπορεί να φαίνονται πολύ εντυπωσιακά, αλλά έχουν να κάνουν ε, με μία συγκεκριμένη περιοχή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχετε κάνει. Φαίνεται ότι έχουμε προοδεύσει πολύ στο θέμα αυτό. Από όλα τα κράτη-μέλη, 15 ήδη ασχολούνται με το θέμα. 14 έχουν αλλάξει τους κανόνες περί ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του γενετήσιου ακροτηριασμού των γυναικών. Ε, ενώ κάποια άλλα έχουν ρητή αναφορά του γενετήσιου ακροτηριασμού στο ποινικό δίκαιο, αλλά απομένουν και κάποια άλλα κράτη-μέλη που δεν αντιμετωπίζουν το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξω τις προσπάθειές σας για επαφές ιδιαίτερα στην Αφρική, αλλά απομένει δουλειά και για μας όσον αφορά ε, το θέμα της δημιουργίας ε, επαφών και της ενημέρωσης εντός της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά το θέμα της ποινική δίωξη. Φαίνεται άσχημο να ασκεί κανείς δίωξη στους γονείς, αν και καταλαβαίνω γιατί θα θέλει να το κάνει κανείς αυτό. Μ' αρέσει πολύ η προσέγγιση σας ε, που επιδεικνύει ευαισθησία απέναντι σε θέματα παραδόσεων. Εάν λοιπόν έχουμε ποινική δίωξη των ε, γονέων ή των ε, άλλων ενόχων εφόσον δεν είναι οι γονείς. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που αν έχουμε τον νόμο δεν θα χρειαστεί να τον εφαρμόσουμε. Αυτό μπορεί να ακούγεται αρνητικό, αλλά φοβάμαι ότι οι ποινικέ διώξει στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι. Ε, μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε, ιδιαίτερα στον κόσμο που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν συμφωνείτε, νομίζω είναι καλύτερο να ακούσουμε άλλες δύο ερωτήσεις και μετά να σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε σε όλες μαζί. Η κυρία Σαπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας πάνω στο θέμα αυτό. Ďakujem Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας στο θέμα αυτό. Είναι η τρίτη μου θητεία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και την πρώτη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό την άκουσα το 2006. Εδώ και 10 χρόνια μιλάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Μιλάμε για τους κινδύνους που ενέχει η πρακτική, καθώς και για την ε, ε, ε, παραβίαση των δικαιωμάτων, την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την διάκριση εις βάρος των γυναικών. Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε με τον αγώνα κατά του γενετήσιου ακροτηριασμού και βλέπετε να υπάρχουν εξελίξεις στον αγώνα αυτό. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια γυναίκες. Ε, δεν ξέρουμε πόσες αναέτος ε, ε, παθαίνουν ακροτηριασμό. Και οι δραστηριότητες σας στην Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία έχουν αποφέρει καρπούς. Νομίζω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει κάνουν πολλά στον τομέα αυτών, αλλά οι πολιτικοί θα πρέπει να κάνουν επίση πολλά. Θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει καλή νομοθεσία κατά του γενετήσιου ακροτηριασμού των γυναικών. Είτε μιλάμε για προληπτική νομοθεσία, είτε για ε, νομοθεσία που να αφορά τις ποινικέ διώξεις, υπάρχουν μεγάλα κενά. Επίσης θα χαιρόμουν αν θα συμμετείχαν περισσότεροι άνδρες στο μέτωπο αυτό κατά του γενετήσιου ακροτηριασμού. Αυτό θα αποτελούσε πολύ σωστό βήμα και θα πρέπει οι πολιτικοί να αναφέρουν πιο συχνά το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. And Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χιμένες, έχει το λόγο, παρακαλώ. Oops. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, ναι, δεν πρέπει να ακούσει Ισπανικά, ναι. Εγώ θα μιλήσω Ισπανικά. Να σα ευχαριστήσω πολύ. Συγγνώμη, αλλά καθυστέρησα. Εγώ είμαι στη δεύτερη θητεία μου. Είμαι πιο πρόσφατη ευρωπούλευτης από την Άννα Ζαμπόρσκα, αλλά παρόλα αυτά έχω αρκετά χρόνια εδώ και από την πρώτη στιγμή από τα θέματα τα οποία προωθώ είναι η αντιμετώπιση των αγροτηριασμών αυτών. Ιδιαίτερα, γενικότερα, η βοήθεια στα θύματα της ε, γενετικής βίας και επίσης και η καταναγκαστική γάμη και τα θύματα καταναγκαστικών γάμων. Και ε, με ενδιαφέρει αυτό που είπατε, ότι ό,τι και να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη, εάν δεν συντονίσουμε τις προσπαθίες μας, αν δεν συνεργαστούμε με τις ε, χώρες προέλευσης, όπου ακριβώς γίνονται αυτοί οι ακροτηριασμοί δεν θα επιτύχουμε σπουδαία πράγματα. Είμαι επίσης μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας. και της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής, ε, Ειρηνικού, όπου συμμετέχουν ε, οι χώρες της Ένωσης και 72 άλλες χώρες, πολλές εκ των οποίων είναι αφρικανικές. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στην Αμίμπια. Εκεί θα συνεδριάσουμε. Σε αυτές μας τις συναντήσεις κάνουμε κάποια προσπάθεια διπλωματικής, κοινοβουλευτικής ε, εργασίας, κάνουμε εκθέσεις με συνεισηγητές από τις χώρες αυτές, επί των οποίων ψηφίζουμε σε αυτές τις συνεδριάσεις. Οπότε έχω συμμετάσχει σε διάφορες τέτοιες συνεδριάσεις, γίνονται μια φορά το χρόνο και πρέπει να αναγνωρίσω ότι ιδίω οι άντρε, ακόμη και μερικέ γυναίκε, ιδίω οι άντρε, πολλέ φορέ λένε ότι είναι τμήμα του πολιτισμού μα. Όταν περνάμε λοιπόν σε ψηφοφορίε για αυτά τα θέματα, υπάρχουν δισταγμοί. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε εκθέσεις, να υποβάλουμε κείμενα διότι σε όσες εκθέσεις κάνουμε για θέματα βίας ε, γενετικής θέτουμε το θέμα των ακροτηριασμών αλλά στην Ευρώπη είναι πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις ξέρω σε κάποιες χώρες είναι κάπως περισσότερες αλλά γενικά είναι λίγες αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι εκεί στις χώρες ε, της Αφρικής οπότε είναι πολύ καλό αυτό που είπατε πρέπει όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις χώρες να το συζητάμε μαζί τους με τις ΜΚΟ, με τους ακτιβιστές εκεί που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Και κάτι άλλο. Ε, πείτε μου αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις χώρες αυτές, για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και όπως ρώτησε και η Άννα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την νοοτροπία, γιατί η νοοτροπία είναι κάτι που δύσκολα αλλάζει γιατί ορισμένοι μπορεί να θεωρούν, ορισμένε γυναίκε μπορεί να θεωρήσουν ότι δεν θα βρουν άντρα, ότι θα είναι λιγότερο ελκυστικέ. Ορισμένοι λένε ότι του αρέσει περισσότερο, για παράδειγμα, στου άνδρε δηλαδή, ο τρόπο που περπατάνε οι γυναίκε που έχουν ακροτηριαστεί. Πρέπει λοιπόν κάπω να αλλάξει η νοοτροπία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο όμω. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις της κυρίας Ότο Γιορτέη. Πολλές είναι οι ερωτήσεις που σας απευθύνθηκαν. Βλέπετε ότι ενδιαφέρονται πολλοί ευρωβουλευτές. Αν γίνεται να μας ενημερώσετε λίγο σύντομα και να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ όσον αφορά το πρώτο ερώτημα που είχε να κάνει με τη δίωξη. Αν πρέπει να ασκήσουμε δίωξη κατά των γονέων. Κοιτάξτε, Τέτοιε διώξει έχουμε δει σε κάποιε χώρε τη Αφρική, δηλαδή γονεί που έχουν υποστεί δίωξη και αν μιλήσετε εκεί με τι τοπικέ κοινότητε θα σα πούνε ότι η δίωξη μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει κατάλληλη ευαισθητοποίηση, αν υπάρχει δηλαδή στήριξη και κατανόηση από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες πολύ συχνά συνειδητοποιούμε ότι δεν έχει γίνει αυτή η απαραίτητη ευαισθητοποίηση, ότι μπορεί να έχει γίνει μια γενική συζήτηση για το ζήτημα. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να ασκήσουμε δίωξη είναι πάρα πολύ σημαντικό η δίωξη αυτή να βασίζεται σε μια πρώτερη ενημέρωση. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό πολλές φορές ήταν προβληματικό. Όταν καταφέραμε όμως να συγκεντρώσουμε τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία, τότε περισσότερες οργανώσεις είπαν ότι όντως θα έπρεπε να προχωρήσουμε τη δίωξη και οι δίωξεις έλαβαν τελικά χώρα. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τις οικογένειες και όσον αφορά κυρίως τα παιδιά και τα κορίτσια, τα οποία πρέπει τελικά να καταθέσουν κατά τον ίδιο των γονέων τους. Αυτό είναι αρκετά προβληματικό, πρέπει να δούμε πώς πρέπει να στηρίξουμε τα κορίτσια αυτά και πώς τελικά δεν θα διαλυθούν οι οικογένειες, δεν θα ταραχθούν οι οικογένειες εξαιτίας της κατάστασης αυτής. Η οργάνωσή μου, η Forward, εργάζεται για το ζήτημα αυτό τελευταία 30 χρόνια. Χρειάστηκαν περίπου 30 χρόνια προκειμένου να καταφέρουμε να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά, ιδίως στα πλαίσια του θεματολογίου για την ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε πιο στρατηγικές προσπάθειες για την καταπολέμηση του κροτεριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτή, μάλλον πάρα πολλοί στο παρελθόν λέγανε ότι δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Τώρα συνειδητοποίησαν βέβαια ότι το θέμα αυτό διαφέρει από τα υπόλοιπα ζητήματα και ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Χρειάστηκε όμως πάρα πολύς χρόνος προκειμένου να αναγνωριστεί το πρόβλημα αυτό, εξίσου με τις υπόλοιπες μορφές βίας κατά των γυναικών. Εξαιτία λοιπόν τη συμβολή των μέσων μαζική ενημέρωση αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό και έχουμε ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι επέρχεται σιγά σιγά μια αλλαγή, υπάρχει μια νέα θετική τάση, η οποία έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που συζητούν το ζήτημα αυτό, υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι οι οποίοι είναι σε θέση να μιλήσουν ανοιχτά για το ζήτημα αυτό και μάλιστα να αναλάβουν και δράση. Και επίσης είδαμε ότι υπάρχει και μία αλλαγή ακόμα και στην ίδια τη στάση των ανδρών, οι οποίοι εμπλέκονται περισσότερο τώρα για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Αρχικά, όταν εργαζόμασταν για το ζήτημα αυτό, δεν είχαμε τη συμμετοχή των ανδρών. Αυτή τη στιγμή, όπω σα είπα, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνδρε, όλο και περισσότεροι πατέρε, οι οποίοι έρχονται και μα λένε, μα αν ήξερα ότι είναι έτσι τα πράγματα, θα είχα λάβει προδειπτική δράση πολύ νωρίτερα. Πολλέ φορέ ακόμα και θρησκευτικοί ηγέτε συντάσσονται μαζί μα. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα σημαντική πρόοδος, αλλά βλέπω ήδη μία πολύ ευίωνη αλλαγή στη στάση των ανθρώπων. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε ανοιχτά για το ζήτημα αυτό και όλο και περισσότερο δίνεται ευκαιρία σε διάφορους παράγοντες να λάβουν δράση προκειμένου να αλλάξει πραγματικά η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να αποφεληθούμε από τη θετική αυτή συγκυρία. Τώρα, έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Ναι, βλέπουμε ήδη ότι υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει μία μείωση στον βαθμό εμφάνισης του φαινομένου αυτού. Ήδη από τα δεδομένα της UNICEF βλέπουμε ότι τα ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου αυτού έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Στην Αίγυπτο είχαμε πολύ ψηλά ποσοστά της τάξης 97%, Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί στο 91%. Τεράστια λοιπόν η μείωση Τη τάξη του 6% όσον αφορά τι γυναίκε που επηρεάζονται από το φαινόμενο αυτό. Χώρε όπως η Κένια από το 30% περάσαμε στο 20-23%. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια θετική αλλαγή. Επίση, ανάμεσα και στα πιο νεαρά κορίτσια, δηλαδή κάτω των 15 ετών, φαίνεται ότι υπάρχει και εκεί μια σημαντική αλλαγή. Υπάρχουν όλο και περισσότερα νεαρά κορίτσια τα οποία δεν υφίστανται πλέον τέτοιο κροτηριασμό. Τα περισσότερα βέβαια δεδομένα βασίζονται σε κάποιες εκτιμήσεις, βασίζονται σε απλά ερωτηματολόγια τα οποία δίνονται σε διάφορους ενδιαφερόμενους. Δεν είναι απαραίτητα αντικειμενικά τα στοιχεία αυτά, πάντως γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να υπάρχουν διαφορετικές μορφές συλλογή δεδομένων, προκειμένου οι εκτιμήσεις αυτές να είναι πιο αντικειμενικές. Και Ασχολούμεθα και με το ζήτημα αυτό, πώς μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εκτίμηση του αριθμού των γυναικών και των κοριτσιών που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό. Τώρα, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με άλλες χώρες, στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας πάντα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ήδη φέτος προσπαθούμε να απευθυνθούμε περισσότερο προς τις χώρες ΑΚΕ, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια σχετική προσπάθεια και ότι προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα το οποίο υπήρχε για το ζήτημα αυτό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Αφρικής. Εστιαζόμαστε όλο και περισσότερο λοιπόν στο ζήτημα του εκτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, νομοθετικά μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα στην Αφρική, όπως ένα σχετικό πρωτόκολλο που έχουμε για τις αφρικανικές χώρες. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τους ανεπτυξιακούς στόχους, όπως ο στόχος 5 αναφέρεται και σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με φαινόμενα όπως ο γενετήσιος ακροτηριασμός. Μια θετική εξέλιξη είδαμε και στον Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Πρωθυπουργό διοργάνωσε μία σύνοδο όσον αφορά το ζήτημα αυτό πριν από δύο χρόνια. Συγκεντρώθηκε πολύ πάρα πολλοί παράγοντες, καταφέραμε να φέρουμε πάρα πολλού υπεύθυνου για τη χάραξη πολιτική, καθώ επίση και εκπροσώπους τη κοινωνία των πολιτών. Μετά την σύνοδο αυτή, μετά τη συνεδρίαση αυτή, είδαμε ότι στα πλαίσια των συζητήσεων πλέον που λαμβάνουν χώρα να λαμβάνεται περισσότερη δράση, ιδίω όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για το ζήτημα αυτό. Εγώ, εργαζόμενοι με κορίτσια, βλέπω όλο και περισσότερο το ζήτημα αυτό προβάλλεται περισσότερο. Χώρε όπω η Γκάμπια. Στις χώρες, στην χώρα εκείνη οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ διστακτικοί να μιλήσουν για το ζήτημα αυτό. Από τότε που ο πρόεδρο τη χώρα όμω μίλησε ανοιχτά για το ζήτημα αυτό και είπε ότι θα το καταπολεμήσει, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρο μιλάει ανοιχτά για την απαγόρευση του φαινομένου αυτού, τότε ξεκινούν πάρα πολλέ προσπάθειε σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσελκύσουμε την προσοχή των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτική σε χώρε όπω η Τανζανία. Είδαμε ότι υπάρχουν πολύ θετικέ αλλαγέ αρχηγοί σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο φυλών συντάσσονται μαζί μας, θρησκευτικοί επίσης ηγέτες συντάσσονται μαζί μας. Είναι σαφές λοιπόν ότι τα πράγματα αλλάζουν, η αλλαγή αυτή μπορεί να είναι αργή πολλές φορές, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε ότι όντως υφίσταται αυτή τη στιγμή μια αλλαγή και ενδεχομένω θα πρέπει να ενθαρρυνθούμε και από τις αλλαγές αυτές και να μην είμαστε πάντα απεσιόδοξοι ακριβώς επειδή η πρακτική αυτή του ακροτηριασμού είναι βαθιά ριζωμένη στην οτροπία των ανθρώπων. Υφίσταται εδώ πέρα και ολόκληρες χιλιετίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι δεν είναι σε θέση να δουν ότι τα πράγματα όντω αλλάζουν. Εγώ όμως βλέπω ότι τα πράγματα αλλάζουν στην πράξη. Στην Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πάντα από 30, πάνω από 30 οργανώσει που μιλάνε για το ζήτημα αυτό. Παλαιότερα ήμασταν η μόνη οργάνωση που δραστηριοποιεί το για την καταπολέμηση αυτού του ακροτηριασμού. Είναι πάρα πολύ εγκαρδιωτικό και ενθαρρυντικό για μένα να βλέπω ότι υπάρχουν όπως και εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαφερθούν για το ζήτημα αυτό. Όσο περισσότεροι είμαστε και όσο περισσότερο μιλάμε για το ζήτημα αυτό και όσο περισσότερο τολμάμε να θέτουμε το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του γενικότερου ζητήματος ε, της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, τότε θα σημειώνουμε συνεχώς πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ήτανε μεγάλη μας χαρά που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Λάβαμε πολλές νέες πληροφορίες και νομίζω ότι η πιο σημαντική Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν ότι μας δώσατε ελπίδα. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας πάνω στο θέμα αυτό και έχουμε επαφή με όλους όσους ε, ασχολούνται με το θέμα αυτό και στην Αφρική και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να λύσουμε το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας είναι στο πλευρό σας, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μας ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστώ και εγώ. so we are going to continue with... Uh, Θα συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Έχουμε την έκθεση με ποιους τρόπους μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ήπεθρο. Έχουμε μαζί μας την ε, συντάκτρια της νομοδότησης, την κυρία Ελίσα Πετκόστιγκερ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Έχω συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μα δίνει η κοινή γεωργική πολιτική για να βελτιώσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο. Εγώ βλέπω το θέμα αυτό ιδιαίτερα από την οπτική των γυναικών. Η γυναική επιχειρηματικότητα στην Ήπεθρο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ιδιαίτερα για την βιώσιμη ανάπτυξη της Ήπεθρου. Στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, το 28% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διευθύνεται από γυναίκες. Σε πολλά κράτη-μέλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50%. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές είναι μικρού και μεσαίους μεγέθους στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο μεγέθους 5,8 εκταρίων. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών όμως ε, εδώ είναι 37%. Όποιος λοιπόν θέλει ίσες ευκαιρίες και για τις γυναίκες ε, θα πρέπει να στηρίξει τις γυναίκες ε, με κατάλληλα μέτρα. Υπάρχουν εδώ λοιπόν κάποιες τέτοιες δυνατότητες. Ζητούμε να υπάρξει υποστήριξη συγκεκριμένα των γυναικών, ε, μεταφορά της γνώσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και μέτρα κατάρτισης, βασικές υπηρεσίες, καθώς και η πρόθεση συγκεκριμένων ε, μοντέλων για την συνεργασία. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ε, που εφαρμόζει πολύ αποτελεσματικά προγράμματα. Έτσι γίνεται πολύ σωστή χρήση των πόρων, μπορούμε όμως ε, και εμείς να συμβάλλουμε στην καλύτερη απορρόφηση των πόρων για να στηρίξουμε όσο γίνεται καλύτερα τις γυναίκες. Πιστεύω, και αυτό αντικατοπτρίστηκε στη γνωμοδότησή μου, ότι θα πρέπει να βασιστούμε περισσότερο σε καινοτόμες ε, μορφές ε, επιχειρήσεων, να έχουμε μέτρα διαφοροποίησης ε, για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Στην πατρίδα μου την Αυστρία υπάρχουν πολλά επιτυχή προγράμματα. Για παράδειγμα, άμεση διάθεση των προϊόντων, όπου οι γυναίκες αναλαμβάνουν την πώληση των προϊόντων στην εκμετάλλευση. Έτσι λοιπόν ε, δεν έχουμε μεσάζοντες στο εμπόριο. Άλλο παράδειγμα είναι ο αγροτουρισμός όπου οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις συνεργάζονται με τουριστικές εταιρείες. Ε, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα παιδιά. Και επίσης έχουμε ε, τον συνδυασμό υπηρεσιών φροντίδας ε, με γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι έχουν την δυνατότητα οι νέες γυναίκες να, ε, να έχουν μια σταδιοδρομία και αυτό είναι καλό και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Θέλουμε λοιπόν ε, συμβουλευτικές εργασίες σχετικά με την ε, διαφοροποίηση, συμβουλές επιχειρηματικές προς τις γυναίκες, καθώς και κατάρτιση. Νομίζω ότι μπορούμε να τα προσφέρουμε όλα αυτά και όλοι ξέρετε ότι έχω χρονικό περιορισμό. πρόβλημα είναι η απορρόφηση των κονδυλίων, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και παροχή συμβουλών καθώς και μείωση της γραφειοκρατίας. Στο σύνολο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ γραφειοκρατία. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Πολύ ευχαρίστω θα λάβω υπόψη μου τις προτάσεις σας. Πρέπει να προστατεύσουμε την ύπεθρό μας, ώστε να παραμείνουν εκεί και οι άνδρες και οι γυναίκες και να μπορέσει να διαμορφωθεί καλά η ύπεθρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα οι σκιώδεις μπορούν να πάρουν το λόγο. Δεν έχουμε εκπρόσωπο των σοσιαλιστών εδώ, αλλά από πλευρά τη ομάδα θα μιλήσει ένας από τους βοηθούς. Παρακαλώ. Θα διαβάσω τη γνώμη της κυρίας Γιώτοβα που είναι η σκιώδης των σοσιαλιστών. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για το σημαντικό αυτό θέμα θα είχε ουσιαστικό ρόλο εάν θέλαμε να υπάρξει ειδικό καθεστώ για τις γυναίκες εντός της ΚΓΠ Στο δεύτερο πυλώνα τη ε, γεωργική πολιτική πρέπει να γίνει ε, περιορισμό κάποιων δαπανών μόνο για τι γυναίκε, Θα βοηθήσει τι γυναίκε στι γεωργικέ ε, και αγροτικέ περιοχέ. Σύμφωνα με μια μελέτη από το Σεπτέμβριο του 2015, οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις χρηματοδοτούνται περισσότερο από το δεύτερο πυλώνα από ότι εκμεταλλεύσεις ε, που τις ε, χειρίζονται οι γυναίκες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ε, βρεφονιπιακοί σταθμοί, σχολεία και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να επιτύχουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Χρειαζόμαστε ειδικού πόρους, περιφραγμένους για να αποφύγουμε την απερίμωση των ε, γεωργικών περιοχών και της υπαίθρου. Και είναι ο ρόλος των γυναικών να παίξουν τον ε, βασικό ρόλο για να το επιτύχουν αυτό και σε εμάς εναπόκειται να τους δώσουμε τα αναγκαία μέτρα και την αναγκαία χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά CCA παρακαλώ, ο κύριος Γκύρικε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ τη Σανθο για αυτή τη γνωμοδότηση Βλέπουμε ότι είναι μια νέα γυναίκα που μιλάει από ίδια πείρα. Καλό αυτό. Να κάνω όμως μερικές συμπληρώσεις που ε, προκύπτουν από συζητήσεις με τις ε, γυναίκες γιοργούς στην περιοχή μου της ε, Πομερανίας και Μέκλεμπουργκ. Μεγάλο ρόλο παίζουν οι μητέρες στη γεωργία που προσπαθούν να συνδυάσουν την επαγγελματική δραστηριότητα με την οικογενειακή ζωή. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τη μητρότητα. Είναι συχνά όμω πρόβλημα η προστασία αυτή. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα, η ε, διαδοχή των γενεών, η, ε, το πέρασμα δηλαδή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τη μία γενιά στην άλλη. Πολλές φορές εγκαταλείπονται πολλές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει να το συνδέσουμε και αυτό. Οι γυναίκες ε, σε ορισμένε περιοχές της υπαίθρου τους ή άλλως σπανίζουν οι περισσότεροι σε βασικές θέσεις είναι άνδρες. Στην ε, ε, Γερμανία μόνο 8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι περίπου 300.000 ε, έχουν ως επικεφαλής γυναίκα. Οι περισσότερες από αυτές μάλιστα υπομερική απασχόληση. Εάν θέλουμε λοιπόν να συνεχιστούν οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις με νέες οικογένειες, τότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν αρκετές γυναίκες για τους ε, άνδρες γεωργούς. Ε, πρέπει να ρυθμίσουμε ό,τι μπορούμε να ρυθμίσουμε. Δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα, αλλά είναι σαφές πρόβλημα και πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο. Κάτι άλλο. Να υπάρχει ασφάλεια για τον προγραμματισμό, ε, για την πώληση των προϊόντων. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα για τα γαλακτοκομικά, αποδεικνύουν ότι πρέπει να εκτιμήσουμε περισσότερο τη δουλειά των γεωργών μας και να αναγνωρίσουμε τη δουλειά αυτή, διότι τους αξίζουν σωστές τιμές και η εκτίμησή μας. Όλα αυτά θα τα συμπεριλάβω σε τροπολογίες προς αυτή τη γνωμοδότηση και προσβλέπω στην καλή συνεργασία για να βοηθήσουμε και τις γυναίκες γεωργούς μας και τη γεωργία μας γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ όμω και ο δισηγητής των Πρασίνων. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την συντάκτηρα τη γνωμοδότηση. Παρακολούθησα το ζήτημα αυτό και στην Επιτροπή Γεωργίας και αποτελεί προφανώ προτεραιότητα για την ομάδα μου. Θεωρούμε ότι η θέση τη συντάκτηρα γνωμοδότηση είναι πολύ θετική, μα δίνει πολλέ ε, χρήσιμε πληροφορίε. Νομίζουμε λοιπόν ότι ε, η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα το βασικό ζήτημα, μάλλον τα βασικότερα ζητήματα περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Ωστόσο, θα θέλαμε να κάνουμε κι εμείς κάποιες προτάσεις οι οποίες θα πάρουν τη μορφή τροπολογιών για να καταφέρουμε να εστιαστούμε σε κάποια διαφορετικά ζητήματα. Πρώτον, έχουμε την διαφοροποιημένη εργασία που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες στην Ήπεθρο είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, ιδίω στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκες που εργάζονται στην Ήπεθρο, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι οι ίδιε ιδιοκτήτε των αγροκτημάτων τα οποία διαχειρίζονται, αλλά εργάζονται για κάποιους άλλους, επιτελώντας όμως την ίδια δουλειά με τους ιδιοκτήτες. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πρόσβαση σε σημαντικέ δημόσιε υπηρεσίε όπω η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση τόσο για του άνδρε όσο και τι γυναίκε. Η εισηγήτρια αναφέρεται στην εξειδικευμένη κατάρτιση. Εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση καταρχά στην γενική εκπαίδευση και παιδεία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, καταρχά. Επίση, κάτι εξίσου σημαντικό για μα και κάτι το οποίο με είχε απασχολήσει και προσωπικά είναι να έχουμε και στις απομακρυσμένες αυτές απομονωμένες περιοχές πρόσβαση σε κάποιες βασικές δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες μεταφορές, παροχή ενέργειας, παροχή διαδικτύου. Εγώ ζω στην Ήπεθρο και όντως δεν υπάρχει καλή σύνδεση με το διαδίκτυο στην περιοχή αυτή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει όμως και με τις δυνατότητε που μου δίνονται να έχω πρόσβαση στο δίκτυο, να μπορώ να δικτυώνομαι κτλ. Πολλά πράγματα εξαρτώνται τελικά από το δυνατό σήμα ή από την καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι εταιρείε παροχή πρόσβαση στο διαδίκτυο υποτίθεται ότι θα πρέπει να καλύπτουν όλη την επικράτεια μια χώρα και όχι μόνο τι περιοχέ εκείνε όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι χρήστε. Και τέλο, και αυτό είναι πάλι εξίσου σημαντικό για μας, και το έχουμε τονίσει σε όλες τις εκθέσεις που έχουμε υποβάλει σε όλες τις επιτροπές, προφανώς θα πρέπει και για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία να τονίσουμε περισσότερο τη διάσταση της ενσωμάτωσης του φύλου, ιδίως για το δεύτερο αυτό πυλώνα στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αυτή τη στιγμή δεν αντικατοπτρίζεται παρκώς στον δεύτερο αυτό πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτέ είναι οι βασικά ιδέε τη δική μου πολιτική ομάδα και είμαι σίγουρο ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε πολύ επικοδομητικά με την εισηγήτρια και εκ πρώτη όψεω είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με, την, με το σχέδιο αυτογνωμοδότησης το οποίο επέβαλε η εισηγήτρια Ακριβώ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε ζουν σε δυσχερεί συνθήκε σε αγροτικέ περιοχέ και περιοχέ υπαίθρου και είναι πολύ σημαντικό για μα να καταδείξουμε ότι οι γυναίκες δεν συνεργάζονται απλώς με τους άνδρες, δεν εργάζονται απλώς στο πλευρό των ανδρών, αλλά ότι και οι ίδιες πολλές φορές εργάζονται, πρέπει να εργάζονται και αυτόνομα. Σας ευχαριστώ πολύ για το κείμενο αυτό. And so, it's the time for the report. Ωραία, μπορεί να απαντήσει η συγγήτρια τώρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά. θα ήθελα να αναφέρω ότι στόχος μας είναι να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις προϋποθέσεις εντός της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σημερίζομαι πολλά, πολλές από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν σχετικά με τα προβλήματα, την προστασία της ε, μητρότητας κλπ. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η κοινωνική πολιτική του κάθε κράτους μέλους ε, όσον αφορά τις ε, συνθήκες στην εκμετάλλευση. Και στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, διαφορετικοί λόγοι που διαφέρει το ποσοστό των γυναικών. Για παράδειγμα, στην Αυστρία συχνά ο άντρας έχει άλλο επάγγελμα και η γυναίκα διευθύνει την ε, αγροτική εκμετάλλευση. Επίσης ε, αναφέρθηκε το θέμα της μητρότητας σε σχέση με τη διεύθυνση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Αυτό συχνά ε, λειτουργεί πολύ καλά στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διότι συχνά η μεγαλύτερη γενιά, οι αγιάδες και οι παππούδες μπορούν να φροντίσουν το παιδί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί παράγοντες εδώ και γι' αυτό συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν, ε, αλλά ε, δεν σχετίζονται απαραίτητα με το ε, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για το οποίο μιλάμε εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβω όλες τις παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του ρόλου των γυναικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν διάφορες επικαλύψεις, τις οποίες όμως ε, πολύ ευχαρίστω θα εξετάσω και θα συμπεριλάβω τις παρατηρήσεις στην γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 30 Μαΐου. Και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών θα πραγματοποιηθεί 9 και 10 Ιουλίου. uh, Προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Ε, διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την εργασία, ε, εγώ δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσω. Ξέρετε ότι έχουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα δώσω όμως το λόγο στην προσκεκλημένη μας. Παρακαλώ.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 Και έτσι προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι η παρουσίαση της μελέτης ε, με τίτλο «Διαφορετικές «Διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την εργασία, την περίθευση και τον ελεύθερο χρόνο». Σήμερα το πρωί είχαμε παρουσίαση και συζήτηση του σχεδίου έκθεσης. Ε, τώρα έχουμε μαζί μας την κυρία Δαβάκη που θα μας παρουσιάσει τη μελέτη. Παρακαλώ. Γεια σας, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πάλι εδώ και που μπορώ να σας μιλήσω για κάποια από τα αγαπημένα μου θέματα που είναι ο συνδυασμός του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου καθώς ε, και τις διάφορες μορφές αδειών. έχετε λάβει όλη τη σχετική μελέτη, η οποία ίσως περιείχε υπερβολικά πολλές πληροφορίες για τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, θα επικεντρωθώ όμως στα βασικά και ελπίζω να μην σας κουράσω πολύ. Βλέπετε εδώ τις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Και έχουμε δύο διαστάσεις, τον χρόνο αφενός και από την άλλη τους πόρους που διαθέτουν οι άντρες και οι γυναίκες. Όσον αφορά λοιπόν την ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, μιλάμε συνήθως ε, για την σχέση ανάμεσα στον ε, δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. Δεν θα μιλήσω για συμφιλίωση ε, εργασίας και οικογένειας, διότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ε, δεν έχουν οικογένεια υπό την στενή έννοια της πυρηνικής οικογένειας. Είναι όμως εξίσου σημαντικό για αυτούς να πετύχουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά τους ε, και ε, την ζωή τους. Σημαντικό είναι λοιπόν να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και η δυνατότητα να μειωθούν ε, οι ώρες ε, εργασίας. Ε, και επικεντρωνόμαστε πάντα στα παιδιά, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Μιλάμε λοιπόν για το spillover effect, όπου υπάρχει όπου πια δεν είναι τόσο καλά διαχωρισμένοι οι τρεις τομείς της ζωής των ανθρώπων. Πρόβλημα είναι επίσης η έλλειψη χρόνου, που είναι η αίσθηση που έχουμε ότι βρισκόμαστε υπό συνεχή πίεση και ότι δεν αρκεί ο χρόνος. Στην μελέτη προσπαθώ να επικεντρωθώ στους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που οδηγούν σε σύγκρουση ανάμεσα στους διάφορους τομείς της ζωής των ανθρώπων. Ε, η οργάνωση του χρόνου ε, έχει να κάνει με την ε, αμοιβούμενη εργασία και την μία αμοιβούμενη εργασία, την εργασία στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη σωστή ισορροπία. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επισημάνω τρεις σημαντικές εξελίξεις. Ε, την στρατηγική 2020 που στόχο έχει ε, να ε, πετύχει 20 εκατομμύρια άνθρωποι να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στη φτώχεια 4,8 εκατομμύρια περισσότερους πολίτες σε σχέση με το 2008. Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 60 ετών ελπίζει να βρει εργασία μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα. Η επιτυχία αυτών των στόχων εξαρτάται από τη λήψη μέτρων καθώς και από την σωστή ισορροπία όσον αφορά τον επαγγελματικό και ιδιωτικό βίο. Κατόπιν έχουμε το Σύμφωνο Ισότητας που τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η σωστή ισορροπία για άντρες και γυναίκες και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ε, εφαρμόσουν οι υπηρεσίε φροντίδα των παιδιών. Και τέλο, έχουμε την ε, στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των δύο φύλων, όπου επαναλαμβάνεται η. η επιμονή για επίτευξη του στόχου για την ε, ισότητα ανδρών και γυναικών στον οικονομικό τομέα, όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, όσον αφορά την μείωση του χάσματος στις αμοιβέ και στις συντάξεις. να εξετάσουμε σύντομα το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν ε, γύρανση του πληθυσμού και ε, αυτό συνδέεται με τις δυνατότητες που δίδονται στις γυναίκες στην ε, αγορά εργασίας. Επίσης, έχουμε επισφαλείς μορφές ε, εργασίας ε, που πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες και σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας που έχουν ε, γίνει πιο έντονες με την οικονομική ύφεση, έχουν οδηγήσει σε τεράστια αύξηση της ανεργίας, επισφαλών μορφών εργασίας, μερικής απασχόλησης και φτώχειας. Οι γυναίκες επίσης ε, παραμένουν ε, οι, ε, κύριοι φροντιστές στις οικογένειες. Έχουμε κάποιες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής 2020 όπου συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική ένταξη των γυναικών. Οι κατευθυντήρες γραμμές του 2020 ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να προωθήσουν ε, την ε, ενεργό γύρανση και τις, να βελτιώσουν τις συνθήκες ε, για αναπήρους νόμους μετανάστες και ευάλωτες ομάδες. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η ισότητα των, των δύο φύλων και μέτρα για την στήριξη ε, γυναικών καθώς και για την ε, μείωση του, της απειλής της ανεργίας. Η φτώχεια είναι σε μεγάλο βαθμό γυναικεία, κάτι που έχει αγνοηθεί μέχρι τώρα. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα πλαίσιο πολιτικής ε, με στοχευμένες πολιτικές. Όσον αφορά τα, ε, τα μοτίβα που βλέπουμε στην ε, απασχόληση, ε, ε, βλέπουμε να υπάρχουν επισφαλείς θέσεις και ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Συχνά υπάρχουν διαφορές και όσον αφορά την αμοιβή, καθώς και τις μορφές των συμβάσεων, καθώς και υπάρχει διαφορά στον χρόνο που δαπανούν στην μη αμοιβούμενη εργασία. Επίσης βλέπουμε σημαντική διαφορά στην ε, σύνταξη που λαμβάνουν άντρες και γυναίκες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απομόνωση των ε, δύο φύλων και βλέπουμε ότι μόνο στο 5% ε, των οικονομικών τομέων υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών ο δημόσιος τομέας είναι πολύ σημαντικός. Ε, βλέπουμε ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται εκεί, ακόμα και στα ανδρικά επαγγέλματα. Επίσης, ε, βλέπουμε υπερεκπροσώπηση των γυναικών ε, στην μερική απασχόληση με θετικές και αρνητικές συνέπειες. Όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας, η μισθή των ανδρών είναι υψηλότερη σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, οι διαφορές ε, όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης ε, δεν είναι τόσο έντονες. Βλέπουμε επίσης ότι η ευμερία των γυναικών που έχουν καταλήψει την ε, αγορά εργασίας είναι χαμηλότερη από αυτές που παραμένουν. Επίσης, οι άντρες εργάζονται κατά μέσο όρο 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες σε 34 ώρες πιο πιθανό είναι οι άνδρες να εργάζονται παραπάνω από 48 ώρες ε, την εβδομάδα. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της εργασίας των γυναικών είναι αόρατο, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή εκτίμηση. Στην παρούσα συζήτηση είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την ισορροπία ανάμεσα ε, στον ε, επαγγελματικό και ιδιωτικό βίο. Έχουμε διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει επαρκή χρήση διαφόρων δυνατοτήτων που γίνονται όσον αφορά την στέγαση της υπηρεσίας κτλ. Ε, τα κριτήρια συχνά δεν είναι σαφή, μπορεί να υπάρχει κοινωνικός στιγματισμός κλπ. Η, σημαντική των, η, σημασία των ε, οικογενειακών πολιτικών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε μια ε, κοινωνία που γυράσκει είναι τεράστια, διότι όλα στρέφονται γύρω από την μη αμοιβούμενη εργασία, τη φροντίδα δηλαδή των μελών της οικογένειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει οριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η φροντίδα είναι μια μορφή εργασίας που έχει πολλές διαστάσεις. Το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται σημαίνει ότι ή είναι πράξη αγάπης, όπου υπάρχει συγγένεια ανάμεσα στον φροντιστή και αυτόν που λαμβάνει τη φροντίδα. Υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συγγένεια, στις οποίες περιπτώσεις πρόκειται για επάγγελμα. Ωστόσο, υπάρχει διαφορά σε σχέση με άλλες μορφές ε, αμοιβούμενης εργασίας, διότι υπάρχει ε, αλληλοεξάρτηση ε, ανάμεσα στα δύο άτομα. Επίσης, υπάρχει κόστος, όχι καθαρά οικονομικό, αλλά και συναισθηματικό. Είτε μιλάμε για τη φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένος. Ο ρόλος πάντα ήταν κυρίως γυναικείος και έχει οδηγήσει σε διάφορες ιδεολογίες. Η παρούσα εικόνα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δείχνει ότι η τεράστια πλειοψηφία ε, φροντίδας παρέχεται από γυναίκες ε, και οι άντρες στερούνται το δικαίωμα να συμμετέχουν εξίσου. Το 2013 οι άντρες εργάζονταν 41 ε, ε, ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες 34 ώρες. Ε, εάν όμως συμπεριλάβουμε την μία αμοιβούμενη εργασία, ε, αλλάζει δραματικά η, η, εικόνα. Εάν συμπεριλάβουμε και τον χρόνο μεταφορές, οι γυναίκ, μεταφοράς, οι γυναίκες εργάζονταν κατά μέσο όρο 64 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι άντρες 53 ε, ώρες. Οι γυναίκες ε, δαπανούσαν 26 ώρες ε, σε μία αμβούμενες δραστηριότητες, ενώ οι άντρες 9 συνολικά. Αυτά είναι στοιχεία του Eurofound 2013. Όσον αφορά λοιπόν τα προγράμματα ενίσχυσης των οικογενειών, μπορεί να λαμβάνουν διάφορες μορφές. Μπορεί να μιλάμε για ε, άμεσες ή έμεσες ε, επιδοτήσεις, ε, άδειε διαφόρων μορφών, πατρότητας, μητρότητας, για εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας κλπ. Μπορεί να έχουμε άμεσες ή έμεσες ενισχύσεις μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ. πολιτικές για προώθηση ε, του συνδυασμού ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου ουσιαστικά ε, βοηθούν ε, στην καθίδρυση του ρόλου του φροντιστή και τίθεται το θέμα εάν οι γυναίκες θα πρέπει να αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την μη αμοιβούμενη εργασία σε σχέση με την αμοιβούμενη. Και είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Ε, στην περίπτωση που οι άντρε επιλέγουν να μην ε, συμμετέχουν ε, στην φροντίδα, περιορίζοντα έτσι τι επιλογέ για τι γυναίκε. Και οι πολιτικές αυτές έχουν να κάνουν και με την οικονομική διάσταση και με την κοινωνική. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή να λάβουμε υπόψη μας τις επιθυμίες εργοδοτών και επιχειρήσεων. Από την άλλη όμως πρέπει να φροντίσουμε και τις οικογένειες. Ε, υπάρχει ε, σύγκρουση όμως ανάμεσα στις δύο αυτές πτυχές ε, όσον αφορά τον χρόνο εργασίας, για παράδειγμα. Τα πακέτα πολιτικής που προκύπτουν από όλη αυτή την κατάσταση συχνά είναι αμφιλεγόμενα το κράτος ε, θα πρέπει να στηρίξει τις οικογένειες ώστε να μην υπάρχει υπερβολικά μεγάλο περιθώριο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Εάν ε, είναι ελάχιστο το ποσοστό της αποζημίωσης σε σχέση με το μισθό, τότε μπορεί κάποιος να επιλέξει πιο σύντομη γονική άδεια. Ενώ εάν υπάρχει θετική σύγκριση ανάμεσα ε, στην αποζημίωση για τη γονική άδεια και τον μισθό, τότε συχνά κάποιος από το ζευγάρι και συνήθως η γυναίκα που έχει πιο χαμηλό μισθό μπορεί να επιλέξει να ε, παρέχει φροντίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει όμως ε, να λάβουμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δηλαδή και το κατά πόσο οι άντρες θα πρέπει να ε, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες για άδεια πατρότητας το θέμα αυτό συνδέεται και με τη μελλοντική σταδιοδρομία της γυναίκας και με το ρόλο του πατέρα. Υπάρχει όμως πάντα ο κίνδυνος απώλειας της θέσης εργασίας, ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι καλές, ή μπορεί να ε, υπάρχει διάκριση εις βάρος ε, των ανθρώπων αυτών από τους εργοδότες. Βλέπουμε η υψηλή χρήση της δυνατότητας ε, γονικής ε, άδεια ε, σε κάποιες χώρες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο χαμηλή η χρήση, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι πολιτικές των διαφόρων χωρών. Μία άλλη πλευρά της παροχής φροντίδας που συνήθως παραμελείται είναι για τους ηλικιωμένους. Αλλά ο πληθυσμός γυράσκει και όλο και περισσότερο. Οπότε χρειαζόμαστε τέτοια φροντίδα και είναι και ηθική υποχρέωση για όλα τα μέλη της οικογένειας, εξαρτήτως φίλου. Και όλοι έχουμε ηλικιωμένους ε, γονείς ή άλλους συγγενείς. 16% των εργαζομένων παρέχουν φροντίδα, 3% πλήρους απασχόλησης και 13% ε, με μερική απασχόληση. Και μεταξύ αυτών που παρέχουν φροντίδα, αυτών που παρέχουν ε, φροντίδα, είναι κατά τέσσερις ποσοστιαίες ε, μονάδες μεγαλύτερε, περισσότερες οι γυναίκες, μεταξύ 18 και 64. τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Αυτά τα στοιχεία όμως δεν αντανακλούν ε, το όρο το τμήμα αυτής της ε, παροχής φροντίδας, γιατί υπάρχουν πολλές άτυπες μορφές παροχής βοήθειας. Είναι πολύ μαύρη αυτή η περιοχή. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι πολλοί που παρέχουν φροντίδα εργάζονται επίσης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ε, άδεια για τα παιδιά για τα παιδιά δηλαδή που πρέπει να φροντίσουν ηλικιωμένους συγγενείς. Και προτείνουν ε, ευέλικτες, ε, ευέλικτα ωράρια, αλλά με χαμηλότερη αμοιβή, άρα δεν είναι πολύ ελκυστικό. Επίσης προτείνονται κάποια φορολογικά ωφέλη για τη συνταξιοδότηση όσων παρέχουν αυτές τις φροντίδες. Η Κομισιόν ε, λέει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διάσταση φύλου αυτό που παρέχουν φροντίδα. Όλοι ξέρουμε θεωρητικά τι σημαίνει αναψυχή. Αλλά αναψυχή ε, μπορούμε να έχουμε όταν κάνουμε όλες τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε, ε, αμοιβόμενες ή όχι. Τι είναι σημαντικό για τη διασκέδαση, την αναψυχή πέρα από το ότι έχει γίνει πολυτέλεια. Είναι λιγότερο επίμαχο, γιατί όλοι ενδιαφερόμεθα για να μπορούμε να διασκεδάσουμε. Αφορά όλες λοιπόν τις κοινωνικές ομάδες, όλα τα επαγγέλματα, αλλά όχι ε, με τον ίδιο τρόπο. Για ορισμένους είναι θέματα επιλογής, είναι θέμα επιλογής. Για άλλους είναι υποχρέωση. Οι δραστηριότητες διασκέδασης ε, παρουσιάζουν επίσης διάσταση φύλου. Επειδή υπάρχουν διαφορές και στις χώρες των 28 όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την απασχόληση, τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε να περνάει να παρισφρεί όλο περισσότερο η εργασία στο χρόνο διασκέδασης. Αλλά η διασκέδαση βοηθάει να μειωθεί το άγχος. Πολλές φορές όμως πρέπει κανείς να μάθει νέες δεξιότητες, ε, να βελτιωθεί γενικότερα. Ε, μία μελέτη του 2013 εξέτασε 46 ευρωπαϊκές χώρες και κατέληξε ότι η σημασία της χαλάρωσης ε, και τη ενασχόλησης με κάτι νέο και διαφορετικό ποικίλει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Αυτοί που είναι πολύ απασχολημένοι ενδιαφέρονται πολύ για να έχουν διασκέδαση. Ενώ οι νέοι και ηλικιωμένοι μαθαίνουν νέε δεξιότητε. Η διάσταση φίλου εδώ είναι η εξής. Πάντα για την, απασχο... για την διασκέδαση. Δεν είναι δικές μου αυτές τις διατυπώσεις. Χρησιμοποιούμε δύο όρους. Τον όρο μόλυνση και κατακαιρματισμός. Δηλαδή η διασκέδαση των γυναικών πολύ συχνά μολύνεται από την παρουσία των παιδιών. Δεν είναι, δεν είναι αρνητική η χρήση του όρου μόλυνση. Όλοι αγαπάμε τα παιδιά. Αλλά οι γυναίκες δεν είναι απόλυτα ελεύθερες να διασκεδάσουν και να απολαύσουν τον ελεύθερο χρόνο τους όπως θέλουν. Ε, βλέπουν ας πούμε τηλεόραση ενώ τα παιδιά παίζουν στο ίδιο δωμάτιο. Η διασκέδαση των γυναικών επιπλέον είναι και πολύ πιο κατακαιρματισμένη από των ανδρών. Και επίση είναι πολύ ενδιαφέρον και το θεσμικό πλαίσιο, γιατί οι γυναίκε έχουν λιγότερο χρόνο για διασκέδαση. Αν λοιπόν δεν αλλάξει η κατανομή εργασία και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, θα παραμείνει αυτή η διαφορά στο χρόνο αναψυχής μεταξύ των φίλων. Σε μια μελέτη της Eurostat του 2015 είδαμε σαφή αρνητική σύνδεση μεταξύ του χρόνου εργασίας, της διάρκειας του χρόνου εργασίας και της ικανοποίησης από το, τη δυνατότητα διασκέδασης. Αυτό απέδειξε ότι στα κράτη-μέλη όπου δαπανώνται περισσότερα για την διασκέδαση και υπάρχει χαμηλότερος χρόνος εργασίας δεν χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ικανοποίηση από τη διασκέδαση. Τώρα τι σχέση έχει αυτός ο συνδυασμός ε, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με την υγεία γιατί είναι απόλυτα σαφές ότι η ευελιξία στον τόπο εργασίας μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Η ευελιξία των ωραρίων. Ακούγεται ωραία ως όρος. Και δίνει δυνατότητα επιλογών στους εργαζόμενους. Αλλά όντως ισχύει αυτό. Είναι τεράστια συζήτηση, δεν θα ασχοληθώ με αυτήν, ε, μη φοβάστε. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί εξετάζοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών για το συνδυασμό προσωπικού επαγγελματικού. Η αύξηση των ευελίκτων των ελαστικών ωραρίων κάνει τη δουλειά να περνάει στον ελεύθερο χρόνο, γιατί οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τηλεεργασία. Άρα δεν υπάρχει χρόνος για να έρθεις ε, σε επαφή με τους ε, συναδέλφους σου στον τόπο εργασίας. Άρα δεν υπάρχει ομαδικό πνεύμα και δεν υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Επίσης ε, η διαίρεση αναφύλω στην εργασία και οι παραδοσιακές επιλογές στον τρόπο ζωής έχουν ως επίπτωση το ότι πολλές γυναίκες σε μεγάλο βαθμό δεν γυμνάζονται δεν έχουν τακτική ε, φυσική δραστηριότητα και αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας. Ένας ε, μεγάλος κίνδυνος με, αυτή, με αυτά τα ελαστικά ωράρια είναι ότι πρέπει συνεχώς να είμαστε στην πρίζα και δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ εργασίας και ελευθέρου χρόνου. Οπότε τέλος, τέλος, Ποιες είναι οι καταληκτικές ε, παρατηρήσεις και προτάσεις πολιτικής της μελέτης. Πρώτη και κυριότερη, αν τα κράτη-μέλη θέλουν να εφαρμόσουν, να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής 2020, οι μακροοικονομικές πολιτικές πρέπει να συνδέονται με κοινωνικούς στόχους. Σε πολλές χώρες η λιτότητα έχει αυξήσει την ε, φτώχεια χωρίς να μειώσει το χρέος, που ήταν υποτίθεται ο στόχος της λιτότητας. Οι μακρονομικές πολιτικές που θέλουν την εξυγίανση, την δημοσιονομική εξυγίανση, πρέπει να βλέπουν τι επιπτώσεις έχουν στην ε, διαφορά αντιμετώπισης των φύλων. Η φτώχεια που είναι πιο υψηλή για τις γυναίκες πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολιστικό τρόπο. Το τονίζω αυτό. Πρέπει η φτώχεια να θεωρηθεί ε, διαρθρωτικό πρόβλημα, όχι ατομικό πρόβλημα. Υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές πολιτικές που μπορούν να μειώσουν την φτώχεια. Για παράδειγμα, το κράτος πρέπει να είναι ο εργοδότης τελευταίας διαφυγής και πρέπει να κάνει επενδύσεις ε, στις ε, φυσικές υποδομές. Οι οικογενειακέ πολιτικές σε περίοδους κρίσης πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και συνεπεί Πρέπει να υπάρχει σωστό συντονισμό και σωστέ διαθροτικές αλλαγέ. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία αυτή. Οι διάφοροι τύποι άδειας μπορεί να βοηθήσουν. Για παράδειγμα, υπηρεσίες ευρωφωνημιακών σταθμών για να μπορούν να εργάζονται οι γυναίκες γιατί η αγορά εργασίας είναι όλο και πιο ανταγωνιστική. Τα σχολεία πρέπει να παρέχουν μετασχολικές υπηρεσίες αλλά και περισσότερη ελαστικότητα στο τόπο εργασίας και διαφορετική τύποι συμβολέων εργασίας. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Η φύση του πακέτου μέτρων και οι δυνατότητες αποζημίωσης πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Πρέπει να έχουμε μία προοπτική για όλη τη διάρκεια της ζωής. Είναι τμήμα των δικαιωμάτων του πολίτη. Νέες μορφές άδειας μπορούν να βοηθήσουν το συνδυασμό μια πολύ καινοτόμα εξέλιξη. Είναι η βελγική πρόβλεψη για διακοπή διαδρομίας Είναι μια άδεια που μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε στη, στη, στη σταδιοδρομία με ένα επίδομα που είναι κάτι ανάμεσα στην αμοιβόμενη και άμυστη εργασία. Η σωστή ισορροπία είναι πολύ βασική Πρέπει να προωθήσουμε την ε, πλήρη εργασία για να αποφύγουμε την ακριβή φροντίδα για τα παιδιά. Με ακούτε? Η κοινωνία των πολιτών πρέπει και αυτή να συμμετάσχει. Η κοινωνία των πολιτών επίσης συμμετέχει στην ε, βοήθεια προς ε, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε διάφορα παραδείγματα στην Πορτογαλία, στην Ανταλουσία, στην Οξφόρδη. το κίνημα αλληλεγγύη για όλους στην Ελλάδα. Ορισμένα μόνο παραδείγματα. Η ποιότητα στην εργασία. Δεν ε, είναι αυτόματα βελτιώσιμη από την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να βοηθήσουμε τα συνδικάτα και τους ε, εργαζόμενους για να αυξηθούν οι μισθοί. Πρέπει επίσης να αλλάξει ο τόπος εργασίας για να αλλάξει και η νοοτροπία προς ε, τις γυναίκες εργαζομένους. Και γενικότερα οι εργαζόμενοι ε, πρέπει να εργάζονται με διαφορετικό, ε, σε διαφορετικό πλαίσιο εργασίας. Οι βραχυπρόθεσμες άδειες μητρότητας δεν είναι αποτελεσματικές. Και τέλος, η ε, ευελιξία και η δυνατότητα να πάρει κανείς τη γονική άδεια κατά τμήματα βοηθάει. Αλλά στην πράξη μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες για τις μητέρες. Αν θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τη μη χρήση αυτών των ωφελημάτων για λόγους ισότητας και καλύτερης ποιότητας ζωής πρέπει να αυξήσουμε αυτούς που μπορούν να λάβουν επιδόματα. Πρέπει να βελτιθούν οι διοικητικές διαδικασίες, να χορηγείται σωστή πληροφορία με σαφή τρόπο, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, να βρούμε τρόπο να ε, απευθυνθούμε σε αυτούς που θα μπορούσαν να ωφελούνται και δεν κάνουν χρήση των ωφελημάτων αυτών. και πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς που αποτελούν όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της ε, Ένωσης, τους μετανάστες, που έχουν σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου για τους πρόσφυγες σε τοπικό επίπεδο για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ε, και υποδομές που χρειάζονται και αυτοί. Ξέρω ότι μία ομοιόμορφη προσέγγιση μπορεί να μην είναι εφικτή λόγω των διαφορετικών πρακτικών και παραδόσεων. Ωστόσο, επειδή είμαστε σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και αύξησης της μετανάστευσης και επειδή η Ευρώπη δεσμεύεται για την ε, ισότητα των φύλων, πρέπει να επιτύχουμε κοινού παρονομαστές. Πρέπει οι πολίτε μα να έχουν αξιοπρεπή επίπεδα ε, διαβίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ κύριε Δαβάκη για την πολύ σημαντική αυτή συμβολή σας στη συζήτηση που κάνουμε όσον αφορά την εξισορρόπηση επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Αναφερθήκατε και σε ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια του ζητήματος αυτού. Αναφερθήκατε στο ότι πρέπει να ισορροπήσουμε την επαγγελματική ζωή με την προσωπική ζωή, με τον ελεύθερο χρόνο. Είναι παρούσα όμως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενδεχομένω να θέλει να πάρει το λόγο για να μας ενημερώσει τη δική της τάση να αφορά αυτά τα ζητήματα. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω και εγώ εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σημαντικότητα αυτή παρουσίαση. Εκτιμούμε πάρα πολύ τα στοιχεία τα οποία μα δώσατε και θα τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά νομίζω ότι μπορούν όντω να μας βοηθήσουν. Με ακούτε. Επί της ουσίας τώρα, οι γενικοί διευθυντές που ήταν σήμερα το πρωί εδώ ανέλησαν εκτενέστατα το ζήτημα αυτό, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. λέω ότι δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είχαμε δύο, γενικές, δύο γενικούς διευθυντές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι εκτενέστατα μίλησαν για το ζήτημα αυτό της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αναφερθήκατε εσείς σε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Εκτιμούμε λοιπόν τη μελέτη σας αυτή και θα την διαβάσουμε πολύ προσεκτικά. Για άλλη μια φορά, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοδομητική σας αυτή εργασία. σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες. Εδαφάκη, αν δεν υπάρχουν λοιπόν ερωτήσεις που δεν υπάρχουν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και προσβλέπουμε βέβαια να λάβουν όλα τα μέλη το έγγραφο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης και το τελευταίο για σήμερα, το σημείο 13 παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Χαρτογράφηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται για τα δικαιώματα των γυναικών σε επιλεγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να κάνω μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό και θα ήθελα να καλέσω εδώ την κυρία Κέιτι Μακ Κράκεν. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή των Γυναικών να λάβει γνώση αυτή τη μελέτη σα για τη χαρτογράφηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με τα φεμινιστικά ζητήματα και ξέρετε ότι θα ή συνεργαζόμαστε και με διάφορες διεθνείς πλατφόρμες οι οποίες απασχολούν και αυτές με τη σειρά τους πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σας ακούμε λοιπόν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη μελέτη αυτή. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική γίνεται στην παρουσίαση μου αυτή είναι και το τέλος της ημέρας. Λοιπόν, εξετάσαμε το πώς λειτουργούν και πώς έχουν τα πράγματα με τις νέες φεμινιστικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούγεται τιτάνιο το έργο αυτό και προφανώς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μια μελέτη που θα κάλυπτε όλες τις νέες φεμινιστικές οργανώσεις. Ανταυτού αυτό το οποίο κάναμε είναι να κάνουμε μία επισκόπηση μιας επιλογής νέων φεμινιστικών οργανώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ένα διεξοδικό, αν θέλετε, χάρτη ή χαρτογράφηση των νέων αυτών οργανώσεων. Θελήσαμε να σας δώσουμε κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα των νέων αυτών μορφών οργανώσεων που έχουν προκύψει τελευταία χρόνια. Να αναφερθώ λοιπόν στα βασικά πορίσματα της μελέτης αυτής Εξετάσαμε 65 οργανώσεις σε 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά τι κάναμε. Προσπαθήσαμε να δούμε τι έγγραφα οι μελέτες έχουν δημοσιεύσει αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, σε ιστοσελίδες για παράδειγμα, ήρθαμε σε επαφή με ορισμένους εργαζόμενους συμμετέχοντε στι μη κυβερνητικέ αυτέ οργανώσει, πάλι βέβαια πάντα ένα μικρό δείγμα, Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα διαφόρων ιδεολογιών σε αυτές τις οργανώσεις όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους τους στόχους. Είναι πάρα πολύ διαφορετικές αυτές οι οργανώσεις. Είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσει κανείς το καθεστώς του νέου φεμινιστικού κινήματος επί του παρόντος, καθότι υφίστανται πολλές διαφορετικές κατακαιρματισμένες ομάδες. Μπορούμε πάντως εν γέννη να πούμε ότι οι νέες φεμινιστικές οργανώσεις, τουλάχιστον αυτές που εμείς εξετάσαμε, είναι πλέον πιο πλουραλιστικές στην προσέγγισή τους σε σχέση με τις οργανώσεις του λεγόμενου δεύτερου φεμινιστικού κύματος δηλαδή της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Οι νέες οργανώσεις τις οποίες μελετήσαμε ασχολούνται πολύ συχνά με το σχετισμό ζητημάτων που αφορούν τη φυλή, τις αναπηρίες, τη σεξουαλικότητα και το φύλλο. Ασχολούνται δηλαδή με, τις, με τα επίμαχα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει σε κάποιους άλλους τομείς και κατά αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται από τους οργανώσεις του λεγόμενου δεύτερου κύματος. Και βέβαια, αυτό το οποίο είδαμε σε όλες αυτές τις οργανώσεις είναι ότι υπάρχει ελάχιστη πρόσβαση σε κρατική κοινοτική χρηματοδότηση. Οι οργανώσεις οποίες εξετάσαμε έχουν σταθεί το πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια. Και οι στόχοι τους είναι ρητός φεμινιστική. Ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών και δραστηριοποιούνται περισσότερο σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια της συζήτησης που λαμβάνει η χώρα σε εθνικό επίπεδο. Επτά χώρες, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάσαμε. Οι περισσότερες από τις οργανώσεις αυτές αν γίνεται την προηγούμενη διαφάνεια να δούμε. Οι περισσότερες λοιπόν από τις οργανώσεις αυτές είναι καταχωρημένες ως μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Πολλές είναι άτυπες οργανώσεις. Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη αν θέλετε. Αναφέρομαι δηλαδή σε οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επίσημη καταχώρηση, κανέναν επίσημο αριθμό μητρώου. Μπορεί να είναι απλά ιστολόγια ή ένα άτυπο διαδικτυακό δίκτυο όπου συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες. Οι οργανώσει αυτέ διαφέρουν πάρα πολύ όσον αφορά τη διάρθρωση του προσωπικού του, Οι περισσότερε βασίζονται στη συμβολή των εθελοντών. Ορισμένε έχουν κάποια διαιτητικά συμβούλια, άλλε πάλι όχι. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη διαφορά προ τη διοικητική του δομή. Και βέβαια τα μέσα κοινωνική δικτύωση και οι επιγραμμικέ πλατφόρμες είναι καθοριστική σημασία για τι νέε αυτέ οργανώσει. Όλε αυτέ οι οργανώσει χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνική δικτύωση για τη δραστηριοποίησή του. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι ε, πολλές από τις οργανώσεις αυτές που εξετάσαμε ανταποκρίνονται με τον ένα τον άλλο τρόπο στις νέες συνθήκες που έχουν προκύψει από τα μέτρα λιτότητας και από την οικονομική κρίση, ακριβώς επειδή στο παρελθόν υπήρχαν επιδόματα ή μέτρα ευνοϊκά για τις γυναίκες, τα οποία δυσανάλογα έχουν περικοπεί και επηρεάζουν αρνητικότατα λοιπόν τις γυναίκες. Αποτέλεσαν λοιπόν νέα αναδυόμενα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται πλέον οι νέες αυτές φεμινιστικές οργανώσεις. Πάρα πολλές μας είπαν ότι προσπαθούν να θεραπεύσουν κάπως τα κακό κείμενα και ότι εστιάζονται στα ζητήματα αυτά κατά προτεραιότητα. Κάναμε κάποιες ε, σύντομες συνεντεύξεις, προσπαθήσαμε να κάνουμε και μια ιστορική ε, ένα ιστορικό απολογισμό του φεμινισμού και το πώς καταλήξαμε σε αυτές τις νέες φεμινιστικές οργανώσεις. Προσπαθήσαμε να δούμε αυτή τη στιγμή αν όντω είμαστε ενώπιον ενό τέταρτου φεμινιστικού κύματος, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τον διαδικτυακό ακτιβισμό, ένα νέο κύμα το οποίο δεν είναι τόσο επίσημο όσο στο παρελθόν, ούτε έχει την κρατική υποστήριξη που είχαν φεμινιστικές οργανώσεις του παρελθόντος. Όπως σας είπα υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά την ιδεολογία που διέπει αυτές τις οργανώσεις. Αν θέλετε ένα κοινό θέμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναλύσαμε είναι ο βαθμός στον οποίο οι νέες αυτές οργανώσεις συνδέονται με τις φεμινιστικές οργανώσεις του δεύτερου κύματος. Ορισμένες από τις νέες λοιπόν αυτές οργανώσεις προσπαθούν να κρατήσουν μια απόσταση ασφαλείας από τις παλαιότερες φεμινιστικές οργανώσεις και είναι πιο ανοιχτές, πιο συμμετοχικές μπορούμε να πούμε σε σχέση με τις παραδοσιακές φεμινιστικές οργανώσεις ιδίως όσον αφορά τον διαχωρισμό των γυναικών ή όσον αφορά των χώρων εκείνων που προβλεπόντουσαν αποκλειστικά για τις γυναίκες, ζητήματα τα οποία προωθούσαν περισσότερο οι παλαιότερες φεμινιστικές οργανώσεις. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν διασυνδέσει απαραίτητα με τι παλαιότερε αυτέ οργανώσει, πάντω οι περισσότερε φεμινιστικέ οργανώσει που εξετάσαμε προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από τις πιο παραδοσιακές φεμινιστικές οργανώσεις. Και κάτι το οποίο ενδεχομένω να σας φανεί λυπηρό είναι ότι ε, οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις εσκεμένα και συνειδητά πέφυγαν τη χρήση του όρου φεμινιστικός ή φεμινισμός, γιατί θεωρούσαν ότι ε, ενδεχομένω να υπάρχει μια αρνητική χρειά πλέον στον όρο αυτό. Μπορούν ότι βέβαια αυτοχαρακτηρίζονται ω φεμινιστικέ, ιδίω στι συνεντεύξει που είχαμε με τα άτομα που, συμμε... που συμμετέχουν σε αυτέ τι οργανώσει και βέβαια καμία από τι οργανώσει αυτέ από και δεν συνδέεται επίσημα με κάποιο πολιτικό κόμμα. Παρακτήσαμε επίσης ότι οι εξεταζόμενες εξεταστήσεις αυτές οργανώσεις ασχολούνται με κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ή με τις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή συγκεκριμένα πλέον ζητήματα, ενώ δεν ασχολούνται τόσο πολύ με μια πιο γενική διαρθρωμένη προσέγγιση του φεμινισμού. Πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν τις νέες αυτές φεμινιστικές οργανώσεις είναι ειδικά ζητήματα, όπως γυναίκες που είναι θύματα ανδρικής βίας, γυναίκες μετανάστες, πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στις επιστήμες, πρόσβαση στις τεχνολογίες, στη μηχανική, στα μαθηματικά, γυναίκες με αναπηρίες, επιπτώσεις των μέτρων της λιτότητας με βάση το φύλλο και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα, την αντίληψη του σώματος ή που έχουν να κάνουν με τον σεξουαλικό στιγματισμό. Πολλές λοιπόν οργανώσεις ήδη στην αποστολή τους, στη βασική τους εντολή μας λέγανε ότι επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και σε συγκεκριμένες ανάγκες προκύπτουν σε αυτές τις ομάδες. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική οργάνωση αυτών των φεμινιστικών οργανώσεων, όσον αφορά την διοικητική τους διάρθρωση, οι περισσότερες είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, χρηματοδότησή τους διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη και η καταχώρησή τους επίσης, η επίσημη διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά οι περισσότερες πάντως, όπως σας είπα, έχουν καταχωρηθεί ως μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και χρηματοδοτούνται όχι μέσω των κυβερνήσεων, αλλά μέσω μονομένων δωρητών ή μέσω χορηγιών. Χορηγιών μπορούν να προκέπτουν και από εταιρείε. Ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πολύ στις συζητήσεις που είχαμε με αυτές τις ε, οργανώσεις. Βέβαια, καθότι δεν υπάρχει επίσημη χρηματοδότηση, βασίζονται οργανώσει οργανώσεις πάρα πολύ στι εθελούσιες δωρεές που γίνονται από μονομένα άτομα ή απασχολούν πολλές φορές προσωπικό με βραχυπρόθεσμες όμως συμβάσεις. Υπάρχουν επίσης διάφορες οργανώσεις που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια ενός σχολείου. Πώς μπορούν, για παράδειγμα, να προωθηθούν κάποια κορίτσια σε κάποιους ε, τομείς που έχουν να κάνουν με τις θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά. Θέλησαμε επίση να δούμε ποια είναι τα εμπόδια αλλά και ευκαιρίε που προκύπτουν ε, με τι ε, νέε αυτέ ε, οργανώσει που, όπω σα είπα, έχουν συσταθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένα σαφέ εμπόδιο, ιδίω στα χρόνια αυτά τη οικονομική κρίση, είναι η χρηματοδότηση, η έλλειψη χρηματοδότηση. Αυτό όμω με τη σειρά του μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία. Πολλέ φεμινιστικέ οργανώσει μα είπαν ότι δεν θέλανε επίσημη κρατική χρηματοδότηση, δεν θέλανε να ενταχθούν με τον ή τον άλλον τρόπο στον κρατικό προπολογισμό, γιατί αυτό τελικά θα τι περιόριζε και ως προς τα θέματα με τα οποία ασχολούνται τους φιλόδοξους στόχους που θέλουν να θέσουν. Επίσης, πολλές οργανώσεις είχαν μια προσέγγιση πολύ πιο αυτόνομη και ανεξάρτητη, προσπαθούσαν να προσελκύσουν περισσότερους εθελοντές, ήταν πιο ανοιχτές προς την ευρύτερη συμμετοχή του κοινού. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει και το ζήτημα αυτό, το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης. Επίσης υπάρχουν αρκετές διαφωνίες και διχόνιες πολλές φορές ανάμεσα στις φεμινιστικές οργανώσεις, ιδίως της Γαλλίας και ανάμεσα σε διαφορετικές ε, γενιές, αν θέλετε, τέτοιων ε, οργανώσεων. Πολλές φορές υπάρχει μια απόσταση πλέον ανάμεσα στους νέους εθελοντές και τους παλαιότερους εθελοντές και αυτό είναι πραγματικά κρίμα και εδώ θεωρούμε ότι χάνεται μια σημαντική ευκαιρία γιατί οι φεμινίστριες των παλαιότερων φεμινιστικών κινημάτων θα μπορούσαν και αυτές να βοηθήσουν τις νέες γενιές. Αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερη πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας και καλύτερη πρόσβαση στους πόρους χρηματοδότησης. Θεωρώ λοιπόν θα μπορούσαν να αποφεληθούν οι νέες αυτές οργανώσεις από τη γνώση και τους πόρους των παλαιότερων οργανώσεων. Επίσης υπάρχει και μια έλλειψη επαγγελματικότητας, αν θέλετε, πολλές φορές και αυτό βάλει κατά της ίδιας της αξιοπιστίας των οργανώσεων αυτών. Κάθε φορά ιδίως που πρέπει να προσελγίσουν πόρους ή επιχορηγήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να φανείς πιστικός όταν εργάζεσαι από την κρεβατοκάμαρά σου, για παράδειγμα. Και είναι πολύ δύσκολο να προσελγίσει κανείς ε, χρηματοδότηση κατά αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, μια ευκαιρία που προκύπτει, αν θέλετε, ένα επίτευγμα των οργανώσεων αυτών, είναι ότι είναι πάρα πολύ προσεκτικές στη χρησιμοποίηση των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένες οργανώσεις έχουν κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκστρατείες που απευθύνονται πάλι σε ένα ευρύτερο κοινό που είχαν πάρα πολύ κάλυψη και στα παραδοσιακά μέσα και που ουσιαστικά κατάφεραν να συμβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο στη συζήτηση για τα φεμινιστικά θέματα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις περιπτώσεις τις οποίες μελετήσαμε, θα προσπαθήσω τώρα πραγματικά να πάω πάρα πολύ γρήγορα. Σας παραθέτουμε εδώ πέρα απλώς στα βασικά μας πορίσματα αναχώρα, στη Βουλγαρία. Καμία από τις εντοπισμένες αυτές οργανώσεις δεν μας είπε ότι είναι φεμινιστική και δεν θέλουν να αυτοχαρακτηρίζουν, να παρουσιάζονται ως φεμινιστικές οργανώσεις. Απλώς ε, υποτίθεται ότι είχαν κάποιους φεμινιστικούς στόχους ή κάποιες φεμινιστικές φιλοδοξίες. Τώρα, αφορά τη Γαλλία. Δεν έχουν τον απαραίτητο προσωπικό, δεν έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση, περισσότερες γαλλικές τέτοιες οργανώσεις και υπάρχει ένας, α, μια ιστορική διχόνοια πολλές φορές και στο πλαίσιο των ίδιων των οργανώσεων. Τώρα στην Ιταλία οι περισσότερες ομάδες προσέγγισης, μάλλον πρόθεσης των στόχο των γυναικών προσπαθούν να εμπλέξουν πλέον και τους άντρες και τις γυναίκες, θεωρούν ότι πάρα πολλά φεμινιστικά πλέον προβλήματα προκύπτουν περισσότερο από τη στάση των ανδρών, άρα θέλουν και αυτούς να τους εμπλέξουν περισσότερο. Δραστοποιούνται περισσότερο με ζητήματα εκπροσώπησης, με ζητήματα κοινωνικής επικοινωνίας, με ζητήματα φιλετικών στερεοτύπων. Όσον αφορά τώρα την Πολωνία, εδώ τα πράγματα επηρεάζονται από το γεγονό ότι η χώρα είναι μια χώρα που έχει προκύψει από ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Πολλές φορές Υπάρχει εδώ πέρα ακόμα μια αρνητική χρειά, η αρνητική προσέγγιση αν θέλετε όσον αφορά τα φεμινιστικά ζητήματα και βέβαια η α, παρούσα κυβέρνηση, το παρόν πολιτικό κλίμα στη χώρα είναι ιδιαίτερα εχθρικό όσον αφορά τα φεμινιστικά ζητήματα. Τώρα στην Πορτογαλία έχουμε μικρές οργανώσεις που βασίζονται κυρίως σε θελοντές και εδώ πάλι είδαμε ότι υπήρχε μια διχόνοια μεταξύ των οργανώσεων αυτών και άλλων ακτιβιστών δεν υπήρχε η απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση ούτε για αυτέ τι οργανώσει. Τώρα όσον αφορά τη Σουηδία. Εδώ πέρα έχουμε μεγαλύτερη διασύνδεση με επίσημα πολιτικά κόμματα, μια καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στη δουλειά που κάνουν αυτέ οι φημανιστικές οργανώσει και άλλοι επίσημοι κρατικοί φορεί για ζητήματα ισότητα και δικαιοσύνη κοινωνική. Στον Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε ότι δεν υπάρχει και εκεί κρατική χρηματοδότηση αλλά εδώ με πολύ πιο ξεκάθαρο τρόπο είδαμε ότι οι φεμινιστικές οργανώσεις δεν επιθυμούν ή δεν χρειάζονται την κρατική χρηματοδότηση. Δεν ξέρω βέβαια αν δεν τους προσφέρεται αυτή η χρηματοδότηση. Πάλι εδώ πέρα βασίζονται πάρα πολύ στη συμμετοχή εθελοντών, έχουν κάποιο έμιστο προσωπικό βέβαια και μας είπαν στον Ηνωμένο Βασίλειο ότι μολονότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα της κοινωνίας απέναντι στις φεμινιστικές οργανώσεις, τα πράγματα τώρα αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση οι ναι, νέες αυτές οργανώσεις δεν θέλουν να παρουσιάζονται, ή να αυτοχαρακτηρίζονται ως αμυγός φεμινιστικές, γιατί αυτό ενδεχομένω να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο που τις βλέπει η κοινωνία. Αυτά είναι συντομία όσον αφορά τη μελέτη μας. Σα ευχαριστώ πολύ. This is Very, how Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει πόσο διαφέρει η κατάσταση από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Υπάρχουν παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Ε, εγώ ίσως έχω μια ερώτηση. Μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι δεν ε, σχετίζονται με πολιτικά κόμματα οι οργανώσεις. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και η ερώτησή μου είναι... Γιατί δεν ε, έχουν εμπιστοσύνη στα διάφορα κινήματα ε, Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας ε, και μάλλον ε, της αξίζει μια ε, πολύ μακροσκελής απάντηση, αλλά η σύντομη απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι οι οργανώσεις έχουν δημιουργηθεί από νέες γυναίκες οι οποίες δεν είχαν επαφή με τις παλαιότερες οργανώσεις και υπήρχε και η επιθυμία από τις νεότερες οργανώσεις ε, να πάρουν απόσταση από τις ιδεολογίες των παλαιότερων. Επίσης, θέλουν να είναι πιο ευρείες οι νέες οργανώσεις, ε, να ε, καλύπτουν ε, διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, ε, διάφορα θέματα που συνδέονται με την σεξουαλικότητα, με την φυλή, την κοινωνική τάξη, την ηλικία κλπ. Το παλαιότερο κύμα φεμινιστικών οργανώσεων επικεντρώνεται περισσότερο σε γυναίκες λευκές της αστικής τάξης. Πρόεδρος, δεν έχω άλλε ερωτήσει. Παρακαλώ. Η κυρία Δαβάκη. Thank you for the... Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το μίσος που περιγράφεται απέναντι στον φεμινισμό. Στη συνεντεύξη σας διαπιστώσατε ότι αυτό συμβαίνει για να έχει κανείς ε, καλή εικόνα στον τύπο ή ξέρουν οι οργανώσεις αυτές ε, τι ακριβώς απορρίπτουν. Ο φεμινισμός ως ιδεολογία είναι τεράστια. Δεν πιστεύω ότι όλα τα μέλη των νέων οργανώσεων, ιδιαίτερα τα νέα μέλη, ξέρουν τι απορρίπτουν. Η κυρία Μακράκεν. Ναι, νομίζω ότι το θέμα αυτό συνδέεται με άγνοια των παλαιότερων ρευμάτων, αλλά μάλλον έχει πιο πολύ να κάνει με την ε, δημόσια εικόνα τους. Ε, δεν θέλουν να συνδέονται με τις ε, αρνητικές χρειές με τις οποίες συνδέεται ο φεμινισμός. Η κυρία Δαβάκη, αυτό όμως ουσιαστικά δεν είναι τελικά εις βάρος ε, των γυναικών και των ε, δικαιωμάτων τους, διότι δεν μπορεί να αποσυνδέσει κανείς τα δικαιώματα των γυναικών από όλους τους κλάδους του φεμινισμού. Και δεν είναι αλήθεια ότι όλες ε, οι πτυχές ε, της φεμιστικής ιδεολογίας είναι οι ίδιες. Ε, παλιότερα είχαμε διάφορους κλάδους. Είχαμε και μαύρες φεμινίστριες. Και νομίζω ότι είναι περίεργο το να είναι κανεί διατομιακό, το να θέλει να είναι μια ευρεία οργάνωση να καλύπτει ε, τόσου ανθρώπου ε, και παρόλα αυτά να απορρίπτουν τον φεμινισμό. Η κυρία και νομίζω ότι απορρίπτουν πιο πολύ τον όρο φεμινισμό, αλλά όταν συνομιλεί κανεί μαζί του, ε, τότε διαπιστώνει ότι αυτό ακριβώ κάνουν. Δεν διαφωνούν απαραίτητα με την ιδεολογία. Είναι καθαρά θέμα δημόσιας εικόνας. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάπως τοξικό θέμα. Διότι δημιουργείται έτσι ένας ε, φαύλος κύκλος ε, σχετικά με την ορολογία. Αλλά αλλάζει η κατάσταση διότι ο φεμινισμός σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο αποδεκτός τώρα που συζητούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι για τα, θέματα αυτά, για τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Μία ακόμα ερώτηση από μένα. Το Κοινοβούλιο τι μπορεί να κάνει ως θεσμικό όργανο όπου εκφράζονται τόσες ε, διαφορετικές ε, ε, απόψεις από την κοινωνία. Ναι, ήθελα να το αναφέρω αυτό. Καταρχάς χρηματοδότηση, αν είναι δυνατόν αυτό. Ιδιαίτερη χρηματοδότηση νέων οργανώσεων επιτρέπουν τη δημιουργία τους και την εκαθίδρυσή τους. Αλλά σημαντικό είναι να ακουστεί και η φωνή των οργανώσεων αυτών και η σημερινή είναι μια πρώτη ευκαιρία να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσει να συνομιλεί κανείς με τις ομάδες αυτές ε, και να ακούει τι έχουν να πούν για τα διάφορα θέματα. Διότι λένε και πράγματα διαφορετικά από αυτά που συζητώνται εδώ μέσα. Σημαντικό είναι λοιπόν να έχει κανείς συνεχή επαφή μαζί τους και να ακούει τις απόψεις τους. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μακράκεν για την εξαιρετική παρουσίασή σας. Και νομίζω ότι το επόμενο θέμα είναι πιο πολύ τεχνικό-διοικητικό. Είναι θέμα για το οποίο απλά θα πρέπει να λάβουν γνώση ε, οι ευρωβουλευτές ε, και η επόμενη συνεδρία είναι στις 30 Ιουνίου. Λήξη της συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ.